των προηγούμενων συνεδριάσεων έχουν διανεμηθεί φαντάζομαι ότι εγκρίνονται εκτός αν ακουστούν αντιρρήσεις μάλιστα είπαμε ότι δεν θα γίνουν τώρα οι ανακοινώσεις της Προέδρου και χαιρετίζω τώρα την παρουσία του Μάριου Ντράγκη η δημόσια αυτή ακρόαση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 109 του κανονισμού του Κοινοβουλίου και είναι τμήμα της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 283 για τον ορισμό των υποψηφίων που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι πρώτες δύο ώρες θα αφιερωθούν σε θέματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον ρόλο της Προεδρίας του Προέδρου της δηλαδή και μετά άλλα 30 λεπτά χωριστά από την ακρόαση αυτή κατά τα οποία θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. ESRB issues, please don't ask it in Λοιπόν, τους πρώτες δύο ώρες επαναλαμβάνω μόνο ΕΚΤ γιατί το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει τέτοιο σαφή διαχωρισμό. Λοιπόν, Χαιρέτησα τους πάντες και πάσες. Θα γίνει τώρα δήλωση του κυρίου Ντράγκη δεκάλεπτη. Μετά οι ερωταπαντήσεις για θέματα ΕΚΤ και μετά ερωταπαντήσεις για θέματα ESRB. Και τέλος τα συμπεράσματα του κυρίου Ντράγκη και εκεί θα τελειώσει το επίσημο τμήμα της συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Μάριο είσαι έτοιμος μάλιστα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Για μένα είναι μεγάλη τιμή η παρουσία μου σήμερα ενώπιόν σας για, στην Επιτροπή δηλαδή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Χαιρετίζω ιδιαίτερα την παρουσία της Προέδρου και όλα τα μέλη που μου δίνουν την ευκαιρία να εκφραστώ εδώ για την αντιμετώπιση των κυρίων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Είναι τιμή μου που είμαι υποψήφιος της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση καθώς και το ευρώ αποτελούν μια επιτυχία που πρέπει να διατηρηθεί προς όφελος όλων των πολιτών μας. Κανένα άλλο πρόσφατο γεγονός, ο συμπεριλαμβανομένης και της κρίσης, δεν μπορεί να αποτελέσει να διαταράξει την επιτυχία αυτή. Τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά. Είπα και πριν ότι είναι τιμή μου η παρουσία μου εδώ στην ακρόασή σας. Φαντάζομαι ότι διαβάσατε το βιογραφικό μου. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τρία πράγματα από αυτού. Η επαγγελματική, την επαγγελματική μου εμπειρία στα δημοσιονομικά, και την αφοσίωση, τη μακροχρόνια μου αφοσίωση στο, στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα υπηρετήσει σε διάφορα τμήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 2006 και ως διοικητής της Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας. Πιστεύω ότι μπορώ να έχω πολύ θετικά αποτελέσματα στην ΕΚΤ παρά το ότι αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και προκλήσεις. Επίσης συμμετέσχον στη λήψη πολλών αποφάσεων που αφορούσαν το ευρώ. Το 1991 ως Γενικός Διευθυντής του Ιταλικού Δημοσίου είχα, ήμουν επικεφαλής της Ιταλικής Αντιπροσωπείας που διαπραγματεύτηκε τη συνθήκη του Μάστριχτ. Μετά συμμετέσχων στη συζήτηση πολλών βημάτων που οδήγησαν στην έγκριση και από την Ιταλία του ευρώ, ιδιαίτερα τις δύσκολες δημοσιονομικές προσαρμογές που χρειάστηκαν στη δεκαετία του 90. Έχω με εμπειρία και σε άλλα ευρωπαϊκά βήματα. Αναφέρω ότι από τον Απρίλιο του 2006 ήμουν πρόεδρος του βήματος για την ε, σταθερότητα που αργότερα έγινε το σώμα υπηρεσία για την μονομισματική σταθερότητα. και έχω ξανάρθει εδώ για να εξηγήσω τις εργασίες του οργάνου εκείνου σε εσά. Τώρα θα ήθελα να πω ότι είναι τιμή μου επίσης που είμαι υποψήφιος πρόεδρος της ΕΚΤ, διότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι μεγάλη επιτυχία. Και επαναλαμβάνω ότι και η πρόσφατη κρίση και άλλα γεγονότα δεν αφισβητούν την επιτυχία αυτή. Το ευρώ έχει φανεί ότι είναι αξιόπιστο και σταθερό δυνατό νόμισμα και οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν πετύχει οικονομική ολοκλήρωση. Η σταθερότητα των τιμών είναι ριζωμένη πια. Τα 12 χρόνια ύπαρξης του ευρώ ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κατά μέσον όρο δεν ξεπέρασε το 2% συμφωνώντας απόλυτα με τον ορισμό της σταθερότητας που είχε θέσει η ΕΚΤ και το Συμβούλιο. Η επιτυχία αυτή είναι σημαντική αν σκεφτούμε σε τι διαταράξεις υπευλήθη η ζωή της Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το χαμηλό πληθωρισμό δηλαδή το λέω γνωρίζοντας ότι έχουν υπάρξει και άλλα ωφέλη από αυτό Χάρη στην αξιοπιστία που κερδίθηκε τα χρόνια αυτά, παρέμειναν σταθε... παρέμεινε σταθερός ο πληθωρισμός παρά την κρίση και παρά την ευελιξία που χρειάστηκε να επιδείξουμε μπροστά σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες. Χωρίς το ευρώ δεν θα μπορούσε να είχε υπάρξει τόσο γρήγορη ανταπόκριση, ούτε τόσο καλός συντονισμός στα νομισματικά. Η αξιοπιστία αυτή πρέπει να διατηρηθεί και πιστεύω απόλυτα σε αυτήν. Νομίζω ότι βασίζεται στην ανεξαρτησία που δίνει η συνθήκη στην ΕΚΤ ώστε να μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόσει την εντολή της, της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών. Επίσης πιστεύω ακράδαντα ότι ως αντιστάθμισμα για την ανεξαρτησία της πρέπει να διασφαλίζει η ΕΚΤ ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων της θα υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια. Καταρχήν προς τους πολίτες και έπειτα προς τους εκλεγμένους ή εκλελεγμένους εκπροσώπους τους. Προσβλέπω στην συνέχιση ενός τέτοιου ανοιχτού και συνεχούς διαλόγου με το Κοινοβούλιο. Με βάση λοιπόν την νομισματική πολιτική καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι η αξιοπιστία που κερδίσαμε δεν θα διαρκέσει αναγκαστικά για πάντα, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Μια σημαντική πρόκληση για την ΕΚΤ είναι πώς θα διαχειριστεί την έξοδο από την τελευταία κρίση και την προοδευτική κατάργηση των προηγουμένων μέτρων της προηγουμένης περίοδου που ήταν απαραίτητα για να υπάρξει σταθεροποίηση και να διατηρηθούν οι ροές των κεφαλαίων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Εμείς, η τράπεζα δηλαδή, στήριξε τη γενικότερη οικονομία της Ένωσης και συνέχισε να διασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών και άρα στήριξε ολόκληρη την οικονομία, αλλά τα μέτρα αυτά και από την ίδια τους τη φύση είναι προσωρινά. έχουν φανεί μια ομαλοποίηση σε πολλές οικονομίες χωρών μελών αλλά και γι' αυτό χρειάστηκε να περιοριστούν οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ. Όμως η ανησυχία διατηρείται από την κοινή γνώμη πολλών χωρών για την κρίση του τραπεζικού τομέα και πολλές τράπεζες εξαρτώνται αυτή τη στιγμή από τη ρευστότητα που μπορεί να εγγυηθεί η κεντρική. Η ασάφεια και η ανησυχία που υπάρχει για τα δημοσιονομικά γενικότερα απαιτεί μια προσεκτική ανάλυση του τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει σιγά σιγά τα έκτακτα μέτρα να καταργηθούν εφόσον δεν χρειάζονται πλέον. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ρευστότητα και η στήριξη της οικονομίας θα διατηρηθεί όσο χρειάζεται. Επίσης όμως να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να λύσουμε τις μελλοντικές ανισορροπίες με τέτοια πάντοτε μέτρα. Ταυτόχρονα ο καθορισμός των επιτοκίων πρέπει να καθορίζεται με βάση την εντολή που έχει η ΕΚΤ, δηλαδή κυρίως τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, για να αποφευχθούν για να αποφευθεί η χειροτέρεψη των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Ούτε η κρίση του χρέους, ούτε η κρίση της ρευστότητας σε ορισμένες τράπεζες δεν μπορούν να αποτρέψουν την έκτα από τη συνέχιση της επίτευξη του κυρίου της στόχου. Δεύτερον, οι προκλήσεις προς την νομισματική πολιτική είναι προκλήσεις δημοσιονομικής σταθερότητας. Η κρίση έθεσε πολλά ερωτήματα ως προς τη σχέση που πρέπει να έχει η Κεντρική Τράπεζα με την νομισματική πολιτική και φάνηκε ότι χρειάζεται περισσότερη διάδραση μεταξύ μικρό και μάκρο οικονομικών μέτρων. Και επίσης έδειξε ότι δεν υπάρχει πραγματική έκπτωση στους στόχους μας λόγω της στήριξης που μπορούμε να δώσουμε σε ορισμένους τομείς. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τη συνέργεια που υπάρχει μεταξύ του δύο τύπων, των δύο τύπων μέτρων, αλλά δεν ταυτίζονται. Η νομισματική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να τονίζει τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα τα ωφέλη από αυτή τη σταθερότητα είναι περισσότερο και όχι λιγότερο φανερά μετά την κρίση. Επίσης, η επιτήρηση των ανισοτήτων είναι κάτι σημαντικό για να έχουμε μία σταθερή νομισματική πολιτική. Επίσης, ο στόχος μας πρέπει να είναι ο μεσοπρόθεσμος ορίζοντας και η ΕΚΤ καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό να τα επιτύχει όλα αυτά, αλλά η νομισματική πολιτική δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο όργανο για να αντιμετωπιστούν αυτά. Η χρήση των λεγόμενων macroprudential εργαλείων μπορεί να είναι καταλληλότερο εργαλείο. Οι νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές μπορούν και αυτές να συμβάλλουν. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η ΕΚΤ παίζει σημαντικό ρόλο και στην ESRB που τις χορηγεί λογιστική και διοικητική βοήθεια. Κατάλληλη διαχείριση της διάδρασης μεταξύ μακροπρουντένσιαλ και άλλων πολιτικών θα ήταν ζωτική. γιατί έτσι μπορεί να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα τεθεί από την διαχείριση της σύνδεσης των δύο τομέων. Σίγουρα είναι σημαντικό να υπάρξει διάλογος μεταξύ των δύο τομέων. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω τις προκλήσεις της οικοδόμησης της ίδιας της Ευρώπης. Το πρόβλημα του χρέους είναι μια πραγματική δοκιμή της ε, σταθερότητας της ίδιας της Ευρώπης και της πολιτικής θέλησης που θα δούμε αν θέλει να επιδείξει η Ευρώπη για να διασφαλίσει την οικονομική της ολοκλήρωση. Η ευρωπαϊκή επιτήρηση των ε, εθνικών προϋπολογισμών απεδείχθη ανεπαρκής. Για πολύ καιρό ε, θετικές δημοσιονομικές συνθήκες έκρυψαν το πρόβλημα που είχαν πολλές χώρες ως προς την οικονομική τους πολιτική γιατί δεν υπήρχαν κοινοί δεσμευτικοί κανόνες η γενικότερη κρίση τόνισε ιδιαίτερα προς τους επενδυτές ότι υπάρχουν κίνδυνοι και αδυναμίες στην αρχιτεκτονική της οικοδόμηση της Ευρώπης και η ανταπόκριση των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών μείωσε τους κινδύνους διάδοσης της κρίσης και διασφάλισε τη σταθερότητα. Η δημοσιονομική στήριξη των χωρών με τα μεγαλύτερα προβλήματα τους επέτρεψε να προσαρμοστούν και να μην καταποντιστούν από τις αγορές. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι το μόνο μέσο. Είναι ένα έκτακτο μέτρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρακάμψεις. Η ανταπόκριση προς το πρόβλημα του χρέους έγκυται κυρίως στην εθνική πολιτική. Σε πλήρη εφαρμογή των σχεδίων προσαρμογής που έχουν συμφωνηθεί. Η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών πρέπει να συνοδεύεται από αίσθημα ευθύνης και συμφωνίας εφαρμογής των κοινών κανόνων. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες αυτές είναι σημαντικά. Οι προτάσεις της καινούργιας Επιτροπής και του Συμβουλίου θα μπορούσαν να είναι και πιο σημαντικά μέτρα, πιο φιλόδοξα για να προφυλαχθούν οι χώρες από τις διαταραχές. Η επέκταση των κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο με, σε αναλογία με τους κανόνες που ισχύουν για κάθε χώρα και ο έλεγχος των εξωτερικών λογαριασμών κάθε χώρας είναι επίσης κάτι θετικό και πάνω απ' όλα οι δομικές αλλαγές που θα στόχευαν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της κάθε οικονομίας πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Όχι μόνο για τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση του χρέους. Γιατί τελικά το μέτρο της επιτυχίας μας θα είναι κατά πόσον μπορούμε να παραγάγουμε ή να προαγάγουμε την ανάπτυξη Πολλά από αυτά τα θέματα βέβαια δεν είναι άμεση ευθύνη της ΕΚΤ, αλλά η ΕΚΤ μπορεί και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να χορηγεί συμβουλές ανεξάρτητες με βάση αξιόπιστα και διαμφισβήτητα στοιχεία. Ελπίζω κατά την ανταλλαγή απόψεών μας να συνεχίσει αυτή η συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση εκ μέρους του ΕΛΚ, ο Ζαν Πολ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, λέει σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας. Θα υποστείτε εδώ Ξαναλέω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε θα υποστείτε εδώ ολόκληρη ανάκριση αλλά δεν θα χρησιμοποιήσω πολύπλοκη γλώσσα για να θέσω τα ερωτήματά μου γιατί είναι απλά καθεαυτά αν και μπορεί η απάντησή τους να είναι δύσκολη. Ο Γερμανός Υπουργό Οικονομικών κ. Σόιμπλε ζητάει αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους μέσα στα πλαίσια του νέου σχεδίου για τη χώρα αυτή. Θέλει τα ελληνικά ομόλογα επίσης και οι ελληνικές τράπεζες να συμμετάσχουν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είπε ότι διαφωνεί με την αναδιάρθρωση αυτή φοβούμενη ότι οι αγορές θα ερμηνεύσουν κάτι τέτοιο σαν νέα έλλειψη ευθύνης των Αθηνών και ότι μπορεί αυτό να θέσει προβλήματα και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Η Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν ε, σε εθελούσια βάση νέα δάνεια. Το θεωρώτημά μου λοιπόν είναι απλό κύριε Πρόεδρε. Αν ήσασταν σήμερα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, ποια θέση θα παίρνατε και για ποιο λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκοζέ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή βέβαια είναι και η σημαντικότερη ερώτηση ε, αυτή τη στιγμή τα πάντα διακυβεύονται γύρω από αυτήν. Όπω πολύ καλά γνωρίζετε, η ΕΚΤ έχει τοποθετηθεί απερίφραστα επί του θέματο. και εγώ συμμερίζομαι την άποψη τη ΕΚΤ και παραθέτω. Η ΕΚΤ δεν είναι υπέρ τη αναδιάρθρωση ή των περίφημων haircuts. Πρέπει να αποκλείσουμε οτιδήποτε δεν είναι προαιρετικό, οτιδήποτε μπορεί να ενέχει το στοιχείο τη ε, υποχρέωση. Θέλουμε να αποφύγουμε την περίπτωση του πιστοτικού γεγονότο ε, και των ε, επιλεκτών ή των γενικών defaults ε, των πτωχεύσεων. Τέλος της παράθεσης. Άρα δηλαδή αυτό που επικρατεί ως άποψη είναι ότι το κόστος ε, της ε, στάσης πληρωμών ξεπερνάει, θα ξεπερνούσε τα ωφέλη. Επιπλέον η στάση πληρωμών δεν θα άγγιζε τα αίτια της κρίσης δημόσιου χρέους. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να καταστήσω σαφές το εξής. Πρώτον, τι είναι ακριβώς αυτό που ορίζουμε ως default. Default στάση πληρωμών θέλετε, αφήνει ανεπίλητα δύο προβλήματα. Εξακολουθεί να υπάρχει πρωτογενέ έλλειμμα το οποίο πρέπει να χρηματοδοτηθεί και μετά τη στάση πληρωμών, μετά το default. Άρα δηλαδή τα χρήματα κάπου πρέπει να ευρεθούν. Οι ε, πολλοί λένε ότι όσοι είναι όσοι είναι υπέρ της στάσης ε, πληρωμών ε, εκ των υστέρων αργότερα θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερο χρήματα. Το δεύτερο θέμα είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες σε μια χώρα που θα κηρύξει στάση πληρωμών αυτοί έχουν τα περισσότερα ομόλογα στα χέρια τους. Επειδή η στάση πληρωμών θα εφαρμοστεί μέσα από haircut αυτές οι τράπεζες θα χάσουν κεφάλαια και κατά πάσα πιθανότητα το κεφάλαιό τους ε, θα εξαφανιστεί πλήρως. Άρα δηλαδή θα πρέπει να βρεθούν περισσότερα κονδύλια για να επανακεφαλαιοποιηθούν οι ε, εσωτερικές τράπεζες. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι σαφές. Αν δεν διατεθούν περισσότερα κονδύλια ή η η φερεγκαιοτητα της χώρας και των τραπεζών που λειτουργούν στην χώρα δεν υπάρχει εγγύηση για αυτές μετά τη στάση πληρωμών, τότε η στάση πληρωμών καθίσταται ε, μια ε, ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία. Άρα δηλαδή αν θέλετε σε γενικές γραμμές το κόστος ε, ξεπερνάει το ωφέλη. Και ας ξαναπάω λίγο πίσω. Γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε την χροκοπία μιας εταιρείας. Μόλις ε, μάθαμε, δεν μάθαμε πλήρως, αλλά μάθαμε πώς να διαχειριζόμαστε και τη στάση πληρωμών μιας τράπεζας. Δεν είμαι και σίγουρος ότι το έχουμε μάθει βέβαια 100%. Αυτό τουλάχιστον για μεγάλες τράπεζες. Δεν έχουμε μάθει 100% όμως πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στάση πληρωμών μιας χώρας. Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όπως σας είπα το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα ωφέλη. Ο κίνδυνος μετάδοσης. Είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε ποια, ποιες είναι οι δίωδοι μετάδοσης ε, που θα προκύψουν μετά από ένα πιστοτικό γεγονός. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, μια άλλη διάσταση του όλου προβλήματος που έχει σχέση ε, με τις στάσεις πλωμών σήμερα και με αυτό που υπήρχε πριν από 10-15 χρόνια. Υπάρχει δηλαδή εδώ σήμερα μια μεγάλη αγορά για τα credit default shops, για τα ασφάλιστρα κινδύνου. Που τι σημαίνει, σημαίνει ότι αν η στάση πλωμών είναι πιστοτικό γεγονός, πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι έχουν στα χέρια τους αυτά τα ασφάλιστρα κινδύνου. Δηλαδή, ποιο έχει ασφαλίσει άλλους κατά της περίπτωσης της περίπτωσης όπου μια χώρα κηρύσσει στάση πλωμών. Μιλάμε για τεράστια ποσά, ως εκ τούτου θα μπορούσε να προκύψει ένα ντόμινο, μια λυσίδα ε, μετάδοση κρίσεων. Πριν λοιπόν τα συζητήσουμε αυτά πολύ συγκεκριμένα, πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία. Δεύτερον, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Μου επιτρέπετε να συνεχίσω για ένα ακόμα λεπτό. Όχι, όχι, δεν έχω άλλο χρόνο. Ίσως μπορεί κάποιος άλλος να θέσει την ερώτηση και θα επανέλθω αργότερα επ' Όχι, αν θέλετε μπορείτε να συζητήσετε για να συνεχίσετε για άλλο ένα λεπτό. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, τίνουμε να υπερτονίζουμε αυτό το θέμα τη αναδιάρθρωση ή τη στάση πλωών. Αν δείτε όμω τι είναι πραγματικά η στάση πλωμών ή η αναδιάρθρωση, είναι κατ' ουσίαν ένας τρόπος χρηματοδότησης ε, τη έκθεση μια χώρας. Γιατί όμως δεν κάνουμε μια διαφορετική ερώτηση. Δηλαδή, γιατί ρωτάμε τι ειναι πραγματικα η σταση πλωμων η η αναδιαρθρωση ειναι κατ ουσιαν ενας τροπος χρηματοδοτησης της εκθεση μια χωρα γιατι ομω δεν κανουμε μια διαφορετικη ερωτηση δηλαδη γιατι ρωταμε τι πρεπει πρωτα απ' όλα να γίνει. Εγώ έχω τη δική μου την προσωπική εμπειρία. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 η Ιταλία ήταν σε χειρότερη θέση από ότι είναι σήμερα η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Τότε δηλαδή είχαμε 11% έλλειμμα του ΑΕΠ και ε, ένα προς 20 ήταν ο λόγος, ο πληθωρισμός ήταν πολύ ψηλότερος, τότε δεν υπήρχε ούτε μηχανισμός ε, του Διεθνούς Δομισματικού Ταμείου, ούτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν κάθε μήνα έπρεπε να εκδίδουμε τεράστιο αριθμό ομολόγων, δηλαδή τριπλάσια περίπου η έκθεση από αυτή που έχει σήμερα η Ελλάδα. Για τρία χρόνια έγινε αυτό. Και το δικό μα το έλλειμμα σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν τριπλάσιο από ό,τι είναι σήμερα τη Ελλάδα. Το 1992 λοιπόν η κυβέρνηση με την συμβουλή τη κεντρική τράπεζα τη Ιταλία ε, εισήγαγε ένα πρόγραμμα το οποίο από τι αγορέ κρίθηκε αξιόπιστο. Χρειαστήκαμε λοιπόν μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά τελικά τα καταφέραμε. Θέλουμε λοιπόν να είμαι απόλυτα σαφή. Δεν υπάρχει ένα εξωτερικό εσωτερικός ε, μηχανισμός. Δεν θα είναι μια ε, μικρή ε, σύντομη διαδικασία. Το 95 τα spread ξεπερνούσαν τις 700 μονάδες βάσης. Είναι αλήθεια ότι μπορούσαμε να υποτιμήσουμε τις, την συναλλαγματική μας τιμία, αλλά μισό λεπτό. Όπως ξέρετε η υποτίμηση είναι ένα ουδέτερο μέτρο εκτός αν παράλληλα προβεί κανείς και σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί μακροπρόθεσμα οι θετικές επιπτώσεις από την υποτίμηση εξαφανίζονται έτσι λοιπόν έγιναν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλάξαμε πάρα πολλά πράγματα όπως ε, παραδείγματος χάνει το μισθολογικό ε, και υπήρξε πραγματική μείωση των μισθών ε, κατά τα χρόνια που ακολούθησαν μετά το 92. Οι ισοτιμίες μπορεί όταν είναι ευέλικτες να είναι και boomerang γιατί, γιατί μπορεί να αυξήσουν τα spread. Έτσι λοιπόν το 95 τα spread τα δικά μας ήταν, εξακολουθούσαν 700 μονάδες βάση σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο ευνοϊκές από ό,τι ήταν κατά τη δεκαετία του 90. Νομίζω λοιπόν ότι ε, πρέπει προσωρινά να, χρησιμοποιήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε κάποια ρευστότητα αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου το κόστος και να νιώθουμε εμπιστοσύνη στο ότι κάτι πραγματικά μπορεί να γίνει. Επόμενη ερώτηση εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών η κυρία Ποντιματά. Μιλήσω ελληνικά κύριε Πρόεδρε. Okay. Θα συνεχίσω στο ίδιο ερώτημα αφού σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας ε, εδώ και θα διευρύνω λίγο το ερώτημα του συναδέλφου του κυρίου Κοζές. Ε, αν σας κατάλαβα καλά από την ε, απάντησή σας, αφήσατε ένα περιθώριο, είπατε δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εσείς αν ήσασταν πρόεδρος σήμερα της ΕΚΤ το ίδιο θα κάνατε, αντιτίθεται κατηγορηματικά σε κάθε ιδέα αναδιάρθρωσης χρέους χώρας μέλους της Ευρωζώνης, ε, εκτός και αν είναι εθελοντική. Ε, ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ε, αυτή η κατηγορηματική αντίθεση περιλαμβάνει και την εθελοντική επιμήκυνση ή την ανταλλαγή ομολόγων που λήγουν με νεότερα στη βάση της πρωτοβουλίας της Βιέννης όπως συζητείτε αυτή την περίοδο και ποιος τελικά θα αξιολογήσει το αν μια αναδιάρθρωση είναι εθελοντική ή όχι, είναι συνάρτηση της ε, ε, απόφασης που θα πάρουν οι τρεις και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για το πότε ερμηνεύεται ε, ότι υπάρχει χρεοκοπία ή όχι. Και με αφορμή αυτό μια γενικότερη πολιτική ερώτηση κύριε Πρόεδρε γιατί έχει σημασία για μας, για τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, αντιτίθεστε έχετε πει και ο ίδιος ότι μια αναδιάρθρωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνέπειες χειρότερες από την κατάρρευση της Lehman Brothers και έχετε δηλώσει και αντίθετος με την εισαγωγή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι το κόστος της κρίσης σήμερα το σηκώνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Πιστεύετε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να αναλάβει ένα μέρος της ευθύνης για την κρίση και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Thank you. Thank you, Madam Podimata. Uh, Madam President, I have a question. Κύριε Πρόεδρε, ήταν δύο ερωτήσεις. Πώς θέλετε να απαντήσω. Έχω έξι λεπτά ή τρία λεπτά. Λοιπόν, ξεκινήστε με την πρώτη ερώτηση. Θα δούμε αν θα φτάσουμε στη δεύτερη. Καταρχήν θέλω να διαβάσω την ε, γραμμή πλεύσεως της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι κατά του κουρέματος ε, αποκλείομαι οποιαδήποτε καταναγκαστική αναδιάρθρωση ε, και υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες. Η μία πρωτοβουλία για μένα είναι τελείως οικειοθελής ε, και η δεύτερη είναι μία για την οποία δεν ήξερα αν είναι ε, θελούσια ή μπορεί να είναι και υποχρεωτική, χωρίς να είναι θελούσια δηλαδή δεν μπορώ εγώ να, κλει, να κρίνω τι γίνεται κυριοθελώς ή όχι γιατί δεν είμαι ε, δικηγόρος αλλά η Λίμαν μας έχει διδάξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί επενδυτές οι οποίοι περιμένουν την ευκαιρία για να υποφεληθούν από τη μη εθελούσια περίπτωση και ε, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να, πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν ε, πολλοί παράγοντες αγορά οι οποίοι με μεγάλη χαρά θα εκμεταλλεύονταν μια κατάσταση ε, άτακτης ή κακο ε, ε, ε, εφαρμοσμένης χρεοκοπίας και αυτό μας έδειξε η περίπτωση της Λίμαν που ήταν η πιο δαπανηρή περίπτωση στην τραπεζική ιστορία και δεν θέλουμε να υπάρξει μία δεύτερη τέτοια εμπειρία. Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται εις την φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Νομίζω ότι απάντησα στο ερώτημα αυτό στο γραπτό ερωτηματολόγιο αλλά ίσως μπορεί να νομίζετε ότι αναφερόμουν μόνο σε νομισματικές συναλλαγές αλλά θεωρώ ότι εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή αυτή η περίπτωση αντιμετωπίζει το ερώτημα κλειδί δηλαδή το ηθικό τον ηθικό κίνδυνο ότι ορισμένα τραπεζικά ε, ιδρύματα έχουν ε, εκμεταλλευτεί την κατάσταση, δημιούργησαν ε, μία ανεξέλεγκτη πορεία η οποία οδήγησε στην κρίση και κατά αυτόν τον τρόπο η κρίση υπήρξε η απόρρια πολλών στοιχείων αλλά αν δούμε ποιοι ήταν οι βασικοί παράγοντες και οι βασικοί παίκτες βλέπουμε ε, πώς ε, διεξήχθη και ε, η φορολογία χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν αναφέρεται στο θέμα αυτό άρα δεν είναι σαφές πώς θα εκάλυπτε ο φόρος αυτός την κατάσταση προς τα έξω και παρόλο που συμμερίζουμε τους στόχους αυτής της φορολογίας έχουμε προβλήματα, προβλήματα εφαρμογής γιατί υπάρχουν δι, τρεις προϋποθέσεις τις οποίες θα θέλαμε να εφαρμόσουμε για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε την ιδέα μιας φορολογίας στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Καταρχήν θα πρέπει να είναι παγκόσμια. Αν δεν είναι παγκόσμια να είστε βέβαιοι ότι όλοι θα προβούν σε συναλλαγές κάπου αλλού ανά τον κόσμο που δεν υπάρχει αυτή η φορολογία. Δεύτερον, εάν διάβασα σωστά τις προτάσεις λέγουν ότι θα είναι βραχυπρόθεσμο μέτρων Πώς λοιπόν θα διακρίνουμε αν πρόκειται για ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο από άλλες πιο μακροπρόθεσμες συναλλαγές και υπάρχουν και διάφορες συναλλαγές βραχυπρόθεσμης διαρκείας. Δηλαδή τα διατραπεζιτικά δάνεια είναι βραχυπρόθεσμα όπως και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τις τράπεζες αλλά όλα αυτά δεν τα θεωρούμε ίσως με από αυτή την οπτική γωνία. Επίσης θέλουμε να αποφύγουμε την κερδοσκοπία. Μπορείτε ε, να εντοπίσετε ακριβώς και να καθορίσετε τι είναι κερδοσκοπία διότι ένα μεγάλο μέρος του hedging ουσιαστικά ε, είναι σαν να προσυπογράφει κανείς ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ε, θα θεωρούμε λοιπόν ότι αυτά είναι κερδοσκοπικές κινήσεις ή και το πιο βασικό είναι ότι οποιαδήποτε φορολογία στα χρηματοπιστωτικά στοιχεία θα θεωρηθεί ότι είναι ε, αρμπιτράζ, μόλχλευση και διατραπεζικές ε, συναλλαγές. Επίσης βλέπουμε ότι όλα αυτά μειώνουν τη ρευστότητα, αυξάνουν ε, το κόστος, ε, αυξάνουν την αστάθεια και είναι προς όφελος των κερδοσκόπων. Εάν λοιπόν πρόκειται για ένα, μια παγκόσμια κίνηση μπορώ να τη δεχθώ και αυτό είναι το γεγονός που θα ήθελα να αναφέρω. Τώρα θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Μόνο μία ερώτηση, διότι χρειάστηκαν επιπλέον τρία λεπτά, άρα κάποιος θα μείνει χαμένος στο τέλος. Εν ονόματι... Ε, η Σιλβή Κουνάρ εν ονόματι της πολιτικής ομάδας. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω εν ονόματι των φιλελευθέρων. Αναλαμβάνετε το έργο σας σε μια δύσκολη εποχή. Τις ερωτήσεις τις έθεσαν ήδη ο Ζωμπόλ Γκοζές και η Άννη Ποδηματά και εδώ θέλω να αναφερθώ στην επικοινωνία. Τεχνικά πιστεύω ότι είστε πολύ ε, έμπειρος και ελπίζω ότι ο καθορισμός σας θα ε, είναι μια νίκη του ευρωπαϊκού πνεύματος επί των ε, εθνικιστικών κινήσεων αλλά ε, ορισμένοι έχουν επιφυλάξεις ε, και σεβόμενος τις γερμανικές αρχές της σταθερότητας της Bundesbank θα θέλαμε να έχουμε κάποιον ο οποίος να βρίσκεται στο κέντρο μεταξύ βορρά και νότου. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσετε την επικοινωνία διότι από πλευράς του Συμβουλίου υπάρχει αποδεδειγμένη κακοποίηση κακοφωνία και θα είσαστε το πλαίσιο αναφοράς για πολλούς Ευρω... Ευρωπαίους ε, θα είστε ο θεματοφύλακας ε, της Ευρώπης ξέρω ότι ο Ζων Κλοντ Κρισιέ έκανε πολλά αλλά πώς θα αναβαθμίσετε την επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς το ευρύ κοινό Ευχαριστώ Ευχαριστώ κυρία Γκουλάρ για αυτή την ερώτηση Ε, είναι δύσκολο να σας πω τι είμαι. Είμαι ένας Ιταλός ουσιαστικά και πολλές γερμανικές εφημερίδες μέχρι ε, προτριμήνου ε, θεωρούσαν ότι κάθε Ιταλός είναι κάτι σαν την πίτσα. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είχαν χαρακτηρίσει. Ουσιαστικά όμως αυτό το οποίο έχω πει τελευταία, τους τελευταίους μήνες όποτε μιλώ δημόσια ε, είναι το ίδιο που έλεγα όλη μου τη ζωή. Ε, είμαι υπέρ της σταθερότητας των τιμών ε, και ε, ίσως αυτό οφείλεται σε κάποιον ο οποίος δεν το είχε όταν ήταν νέος ε, στην Ιταλία όπου είχαμε πληθωρισμό πέραν του 20% και ε, όταν εγώ θέλω να υπάρχει φορολογική αναδίπλωση οφείλεται στο ότι πέρασα την δεκαετία του 90 στην Ιταλία δεν είμαι δηλαδή μια αυθεντία έχω πλήρη ευαισθησία προς τους άλλους αλλά ουσιαστικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία θεωρεί ότι η μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλο το χώρο. Ε, δεν υπαγορεύεται από τις εθνικές συνθήκες, τις εθνικές ε, προτεραιότητες ή προτιμήσεις και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σαφές στο μυαλό μου. Δηλαδή, όπως είπα και στην αρχή, είμαι υπόλογο σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και σε και όχι προς τους πολίτες μίας χώρας. Πέραν αυτού όμως θα είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσω τον Ζων Κλωτρισέ στο ύψος του. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς στο ίδιο επίπεδο. Ευχαριστώ υπέρ των Ευρωπαίων Συντηρητικών η κυρία Βίνλετ ο πρόεδρος της, ε, Γιούγκερ ομολόγησε ότι προτιμάει η ECRB ε, να έχει έναν ε, επίσημο ρόλο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρώ αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτό το ρόλο. Θα θέλατε σε ένα ρόλο διαχείρισης και τελικά ε, εάν άλλαζαν οι συνθήκες θα σας προσέφεραν αυτό το ρόλο και αν όχι γιατί όχι. Thank you, Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη αυτή η ερώτηση. Ε, το έχω πει νομίζω επανειλημμένα. Η πρωταρχική εντολή ή εντολή αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, του ε, ECRB του συστήματο του ε, συστημικού ελέγχου είναι να καθορίζει και να διασφαλίζει την σταθερότητα τιμών. Αυτό είναι ο βασικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου. Που σημαίνει ότι δεν είναι καλή ιδέα να εφαρμόζουμε μια νομισματική πολιτική έχοντας κατά νου ένα, μια συγκεκριμένη ισοτιμία στόχο. Αυτό δεν το κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και ούτε και η Ευρωζώνη το πράττει αυτό, αλλά ούτε και εμείς ε, το κάναμε κατ' ουσίαν κάτι τέτοιο. Διότι κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θυσιάζουμε το στόχο της σταθερότητας των τιμών. Ε, εγώ λοιπόν ε, σε αυτή τη φάση αυτό θέλω να πω και νομίζω όλοι είμαστε σαφώς κατά της υπερβολικής διακύμανσης των ισοτιμιών. Όλοι είμαστε υπέρ της σταθερότητας των τιμών, αλλά ο τρόπος για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο είναι σε παγκόσμιο επίπεδο να διασφαλίσουμε ότι δεν προκαλούμε ανισορροπίες σε παγκόσμια επίπεδα με υπερβολικά ελλείμματα ή πλονάσματα των, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών πρέπει να βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση έτσι ώστε να παρεμποδίζονται οι υπερβολικές διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα εξ ονόματος των Πρασίνων, ο κύριος Κάνφα. Καλημέρα. Θα χρειαστείτε τα ακουστικά. Καλώς ήρθατε κύριε Διοικητά. Θα ήθελα να πω κάτι που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα, ούτε από εσά, ούτε από τους υπόλοιπους συναδέλφους, το όνομα Goldman Sachs. Στην παρουσίασή σας περάσατε από τη διοίκηση της Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας στην ευρωπαϊκή σας καριέρα και ξεχάσατε τον καιρό που περάσατε στο Goldman Sachs όπου ήσασταν αντιπρόεδρος υπεύθυνος για την Ευρώπη για τα χρέη συγκεκριμένα. Γνωρίζετε βεβαίως τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ Goldman Sachs και Ελλάδας το 2000. Ο σκοπός μου δεν είναι εδώ να σας επικρίνω, αλλά νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, λόγω της εντολής που ίσως λάβετε του διορισμού σας, θα θέλουν να έχουν εμπιστοσύνη στον προ... μέλλοντα πρόεδρο της ΕΚΤ και θέλουμε εξηγήσει γιατί μέχρι τώρα απαντήσατε μόνον ότι δεν ήταν δική σας δουλειά, δεν ανακατευτήκατε καθόλου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το swap, αυτή η συμφωνία Goldman Sachs και Ελλάδος ναι μεν είναι από το 2002 αλλά η δουλειά σας εκεί ως αντιπροέδρου ήταν ακριβώς να πουλάτε, να προωθείτε τις εξυπηρετήσεις του Goldman Sachs σε χώρες σαν την Ελλάδα. Το 2003 ήσασταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με μία συνάδελφο Ελληνίδα η οποία ακριβώς χειρίστηκε αυτή τη συμφωνία του ΣΟΑΠ. Τι έχετε να μας πείτε λοιπόν σήμερα παραπάνω από αυτά που είχατε πει σε μία σύντομη δήλωση που έλεγε ότι απλώς δεν είχατε καμία σχέση και που μου φαίνεται λανθασμένη. Well, I mean, if you already know it's not the truth, αν ήδη γνωρίζετε την αλήθεια, γιατί ρωτάτε. Ας απαντήσω, τέλος πάντων. Είναι σημαντική ερώτηση και σας ευχαριστώ που τη θέσατε. Αν βεβαίως σας ικανοποιήσει η απάντηση. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να έχει δράσει κανείς με ακαιρεότητα, αλλά και να είχε σκοπό την ακαιρεότητα. Uh, Goldman Sachs. Uh, Πρώτον, η εμπειρία μου στον Goldman Sachs. Οι συμφωνίες Goldman Sachs και ελληνικής κυβέρνησης είχαν αναλυφθεί πριν να πάω εγώ στον Goldman Sachs. Αυτό το έχω πει ξανά και ξανά. Δεύτερον, δεν είχα καμία σχέση με τις συμφωνίες αυτές. Τρίτον, νομίζω ότι οι πληροφορίες σας δεν είναι απολύτως ακριβείς. Δεν ήμουν υπεύθυνο προώθησης συμφωνιών σε κυβερνήσεις. Εγώ συνεργαζόμουν με τον ιδιωτικό τομέα και αν και ο Goldman Sachs ήθελε να συνεργάζομαι και με το δημόσιο τομέα, εγώ τους είπα ότι επειδή τον ξέρω το δημόσιο τομέα δεν έχω κανένα ενδιαφέρον, δεν θέλω καθόλου να συνεργάζομαι με τον δημόσιο τομέα. Και στο τέλος της θητείας μου εκεί κατά το 2005 με ρώτησαν αν πάλι θέλω να αναλάβω τον δημόσιο τομέα και δεν έγινε τίποτα ούτε τότε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα για αυτές τις συμφωνίες, ούτε έκανα τίποτε αργότερα ή πριν σε σχέση με τέτοιες συμφωνίες. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Πάντα μπορεί κανείς να πει ότι ε, αφού ήσουν με τις επενδυτικές τράπεζες συμφωνούσατε και μαζί τους. Δεν είχατε κα... μήπως ε, αντιτιθέμενα συμφέροντα. Εγώ ως διοικητής Ιταλικής Τράπεζας έχω αποδείξει ότι δεν υπήρξε τίποτα τέτοιο. Μάλιστα. λόγω της επιτήρησης που κάνει η Banca d'Italia γνωρίζουμε ότι καμία Ιταλική τράπεζα δεν είχε πρόβλημα κατά την κρίση. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά ένας είναι αυτή η επιτήρηση. Και ίσως είναι και μοναδική η περίπτωση αυτή της Ιταλίας. Μήπως ήμουν υπερβολικά καλός με τους Ιταλούς τραπεζίτες, ρωτήστε τους. Θα μπορούσε πάντως κανείς να πει ότι στο κάτω-κάτω well, το βήμα, το φόρουμ της σταθερότητας ούτε εκεί μπορεί κανείς να πει ότι ήμουν υπερβολικά μαλακός. Αυτά που λέει το FSB για την κρίση θα ξέρουμε από το 2002 μπορώ να σας στείλω την παραπομπή εκεί διετύπωσα πολλές προειδοποιήσεις για τον επερχόμενο κίνδυνο μαζί με τον καθηγητή Τζαβάτσι και τον καθηγητή Μέρτον. Να, διαβάστε εδώ. Εδώ αναλύουμε καταστάσεις όπου αναμένονται απρόσμενοι κίνδυνοι, συσσωρευμένοι ιδιαίτερα τις εγγυήσει που δίνουν οι κυβερνήσεις σε τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που μπορεί να καταλήξουν στη συσσόρευση απρόσμενων κινδύνων για την εξισορρόπηση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και συνεχίζει έτσι. Από ό,τι ξέρω αυτή είναι η πρώτη συζήτηση των ΣΥΦΙΣ που λέμε. Υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις στον τύπο όταν προείδρευα της FSB για προειδοποιήσεις. Αν επειδή είχα δουλέψει στον Goldman Sachs τα έλεγα όλα αυτά δεν το ξέρω αλλά δεν νομίζω. τελική απόδειξη είναι ότι αυτά που πράξαμε στο FSB ως τραπεζικές διευθετήσεις. Το 2008 η μόνη ανταπόκριση στην κρίση δόθηκε από τις 77 συστάσεις που έγραψε η FSB. Αυξήθηκε το κεφάλαιο τραπεζών σε επίπεδο που δεν το ανέμεναν καν. Υπήρξε η Βασιλεία 3, υπήρξε η συζήτηση των ΣΥΦΙΣ και άλλα, αλλά ας σταματήσω εδώ και ελπίζω να σας έχω πείσει. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν ο κύριος Γιούγκεν Κρουτ εκ μέρους της ε, Γκουε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Ντράγκη, ε, θα ήθελα μισό λεπτό αν έχετε καλοσύνη να περιμένετε για τα ακουστικά. Κύριε Ντράγκη, σας ε, καλωσορίζω θερμά και εγώ θα ήθελα να συνεχίσω με αυτή την ερώτηση ε, επί της οποίας απαντήσατε εν μέρη. Θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής ότι στις εφημερίδες που διάβασα στη Γερμανία ε, κανείς ε, δεν αμφισβητεί την τεχνογνωσία σας, τις γνώσεις σας. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση κυρίως σε σχέση με τη μελλοντική σας θέση. Όμως υπάρχει αυτή η πολιτική αχίλιος φτέρνα για την Goldman Sachs και για την Ελλάδα. Ακόμα και δεν είναι πλακήκατε σε αυτή την περίπτωση, παρόλα αυτά ε, παραμένει το γεγονός ότι εσείς δουλέψατε σε ένα πλαίσιο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Μια γερμανική εφημερίδα ε, αναφέρει ότι μένει έτσι μια πικρή γεύση από αυτό το γεγονός. Γνωρίζετε την κατάσταση στην Ελλάδα, στην Ιταλία, ε, στην Ισπανία. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι στους δρόμους, υπάρχουν πολλές αναταροχέ. Γι' αυτό λοιπόν αν θέλετε έχοντας σε αυτά κατά νου να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά το καθήκον σα, κυρίω σε σχέση με την Ελλάδα, πρέπει να χαρακτηρίζεστε από ιδιαίτερη ακαιρεότητα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ιστορία με την Goldman Sachs αποδυναμώνει την αξιοπιστία σα για το μελλοντικό σα ρόλο. Και γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό που ρώτησε και ο Πασκάλ. Δηλαδή την απαραίτητη αξιοπιστία, έχοντα κατά νου όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, Πώ σκοπεύετε να την επαναφέρετε. σα ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η απάντηση που έδωσα προηγουμένως είναι κατ' ουσίαν η απάντηση στην ερώτησή σας. Δηλαδή, εγώ νομίζω, είπα, ότι λειτουργήσα με ακαιρεότητα και θεωρώ ότι αυτό μπορούν να το κρίνουν ε, και όσοι είναι αμερόληπτοι. Ε, θα καταλήξουν ότι όσο ήμουν στην Goldman Sachs ήμουν πραγματικά ακέραιος και αμερόληπτος. Και νομίζω έχω καταθέσει πάρα πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ε, παρουσία μου στον ιδιωτικό τομέα και στη συγκεκριμένη αυτή τράπεζα όταν ήμουν εκεί επουδενή δεν βοήθησα, δεν προτίμησα τις ε, εγχώριες ε, τράπεζες της Ιταλίας για τις οποίες ήμουν αρμόδιος ε, σε θέση επόπτου. Κάθε άλλο μάλιστα. Ήμουν σκληρός απέναντί τους και στην της d'Italia έτσι κι αλλιώς όσοι εργάζονται εκεί πιστεύουν ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να ασκεί κανεί τα εποπτικά του καθήκοντα. Ανεξάρτητος, με υπευθυνότητα, με αυστηρό έλεγχο. Στις δημόσιες δηλώσεις που έχω κάνει έχω αναφέρει πάρα πολλά στοιχεία για τους κινδύνους που είχα διαβλέψει, που σωρεύονταν ήδη τότε και αυτό το είπα με την ιδιότητά μου ε, του Προέδρου ε, του ε, του FSB, του Financial Stability Board. Και είχα πει και είχα αποδείξει ότι οποτεδήποτε είχα αρμοδιότητες ρυθμιστικές απέδειξα ότι θα χρησιμοποιούσα αυτές τις αρμοδιότητες μου για να υπάρχει ένα καλύτερο σύστημα για το μέλλον, πιο ανθεκτικό. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να έχω κάνει ή τι θα έπρεπε να απαντήσω στην ερώτησή σας. Νομίζω ότι αυτά που είπα αποτελούν από μόνα τους την απάντηση. Ωραία. Και τώρα ο Μάριο Μποργέζιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι αυτές οι δύο τελευταίες ερωτήσεις ε, κατά κάποιον τρόπο εισήγαγαν ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή μου είναι γενικότερο. Αυτό το θέμα της Goldman Sachs ε, κατά την άποψή μου αυτό δημιουργεί κάποιες ε, ανησυχίες ε, σε πολλούς παριστάμενους. Ε, εμείς που συμμετείχαμε στην ΣΟΥΡΕ, στην Επιτροπή Κρίσης, έχουμε ακούσει επανειλημμένα πολλούς να λένε ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για την περίπτωση μια νέα κρηματοδοτική κρίση κάτι που θα ήταν απόλυτη καταστροφή για ορισμένε χώρε μεταξύ των οποίων και η δική μα. Έτσι λοιπόν, κάτω από όλα αυτά και κάτω από αυτό το πρίσμα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό εσεί να ξεκαθαρίσετε ορισμένα πράγματα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι περιβάλλοντα, όπως αυτόν τη Goldman Sachs, αλλά και άλλα συναφή περιβάλλοντα, έχουν σχέσεις ε, με το Λέσχη Μπίλντερμπεκ, σχέσεις ε, με ομίλους πολύ συντηρητικούς. Ε, εσείς λοιπόν εκφραστήκατε ριζικά και κατηγορηματικά απέναντι σε αυτή την πρόταση του να επανευρεθεί ένα σύστημα που θα προβλέπει ξεκάθαρο διαχωρισμό από τις ε, τράπεζες που ασκούν κερδοσκοπία από τις υπόλοιπες. Γιατί υπάρχει έτσι μια συγκεκριμένη άποψη που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κουραστεί πια να πληρώνουν τα χρέη των ε, υψηλών μεγάλων τραπεζών που δανείζονται. Και εγώ τέλος πάντων θέλω να κάνω μια ερώτηση, μια ερώτηση που έγινε και από τον κύριο Ντιπιέτρο από ένα κόμμα με το οποίο εγώ δεν έχω καμία πολύ σχέση, αλλά θα αναφερθώ σε αυτό ε, σε σχέση με τα το οικονομικα Σας ερωτώ λοιπόν, εάν εσείς τελικά αποκτήσετε αυτή τη θέση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συγγνώμη λέει η πρόεδρος, διακόπτη, Μπορείτε να μας ε, ξεκαθαρίσετε τη θέση σας σε σχέση με την νομισματική κυριαρχία των κρατών. Εσείς αναφέρετε σε, αναφέρετε σε διάφορους οργανισμούς ε, και η περιγραφή αυτών των οργανισμών υπάρχει. Αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε και μετά κατηδίαν, αλλά μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο. Είναι οργανισμοί όπου πήγα εγώ, αλλά ήταν και άλλοι πάρα πολλοί Ιταλοί, όπως ο κύριος ε, Τρεμόντι, ο Δόκτωρ Μπερναμπέ και πάρα πολλοί άλλοι. Δεν νομίζω λοιπόν ότι εκεί μιλάμε για μυστικέ μυστικές συμφωνίες. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι οι επενδυτικές τράπεζες ανήκουν ακούν του Μία παρατήρηση εκτός μικροφώνου, Δυστυχώς εμείς δεν την ακούσαμε. Ο κύριος Ντράγκη συνεχίζει λοιπόν. Αυτοί οι οργανισμοί και αυτές οι λέσκες είναι διαφανείς. Ε, δεν είναι μυστικές όπως σας είπα. Τώρα, όσον αφορά αυτόν τον σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε επενδυτικές τράπεζες, trading activities για να το πούμε πιο ξεκάθαρα και άλλες δραστηριότητε των τραπεζών, τον πλήρη διαχωρισμό, εγώ δεν ήμουν ποτέ αντίθετος. Τον αντίον, αυτό είναι ένα κομμάτι του μενού των επιλογών που έχει έχουν προσφερθεί στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αν λοιπόν η Ευρώπη θεωρεί ότι αυτή είναι μια εναλλακτική λύση, βεβαίω και μπορεί να την ακολουθήσει. Είναι η εναλλακτική λύση που έχουν επιλέξει οι Ηνωμένε Πολιτείε. Προφανώ βεβαίω εξαρτάται από την τράπεζα, από τη μορφή τη τράπεζα, αλλά και από τη χώρα όπου λειτουργεί η τράπεζα. Όσον αφορά την νομισματική κυριαρχία, αυτό ρυθμίζεται από τη συνθήκη του Μάστριχ. Έχει τοποθετηθεί από αυτού και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο στόχο είναι πάνω απ' όλα η σταθεροποίηση μέσω μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση των τιμών. Ευχαριστώ. Επανερχόμαστε στον Βέρνερ Λάνιον και στο ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε Ντράγκη, Είστε ένας έμπειρος ειδικό και στη Γερμανία ορισμένοι σας θεωρούν ως τον πλέον κατάλληλο. Θέλω να προσθέσω μία ερώτηση στα σχόλια τα οποία μόλις κάνατε σχετικά με τις ανισορροπίες στην Ευρωζώνη. Είπατε ότι η Ελλάδα δεν είναι στο χάλι της Ιταλίας στη δεκαετία του 90 και η Ιταλία ήταν πολύ μεγάλη μεγαλύτερη χώρα. Αλλά στο θέμα της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωζώνη η η ανταγωνιστικότητα αποκλίνει μεταξύ των χωρών όλο και περισσότερο. Τι προτείνεται λοιπόν για την Ευρωζώνη κατά τρόπον ώστε πέραν της νομισματικής πολιτικής να βελτιώσει κανείς την ανταγωνιστικότητα ιδίως στα κράτη τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Λάνιεν. Αυτό είναι πολύ βασικό ερώτημα, διότι έχει σχέση με την διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής σε μια ετερογενή περιοχή. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι ο στόχος, ο στόχος της ΕΚΤ είναι να έχουμε μέσω πρόθεσμη ε, σταθερότητα τιμών για όλη την περιοχή. Το ερώτημα είναι αυτό θα εμποδίσει τις πιο αδύναμες χώρες εάν αυξηθούν τα επιτόκια ε, για λόγους σταθερότητας των τιμών. Η απάντηση είναι ότι ας κοιτάσουμε ποιο είναι το κόστος του, ε, των πιστώσεων γιατί αυτό είναι το θέμα το οποίο μας απασχολεί και αυτό έχει στενή σχέση με το κόστος ε, των κυριάρχων χρεών διότι όταν οι τράπεζες ε, επενδύουν χρήματα κοιτάζουν τις ενελεκτικές επενδύσεις όταν βλέπουμε μια χώρα που έχει φορολογική κρίση το κόστος ε, του χρέους είναι 14-15% για το κυρίαρχο χρέος και αυτό είναι ε, πολύ υψηλό σε σχέση με ε, τις, ε, τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια της ΕΚΤ. Τι προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι για να εξασφαλίσει κανείς την ε, σταθερότητα των τιμών θα πρέπει να χαμηλώσει όλα ε, τα επιτόκια και για τις χώρες που πάνε καλά και για αυτές που πάνε λιγότερο καλά. Και για να μειώσουμε το κόστος ε, των δανείων πρέπει να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα φορολογικής αναδίπλωσης που θα μειώσει το χρέος αυτό εις ε, το ισχύον δημόσιο χρέος. Η σταθερότητα λοιπόν θα μειώσει τα επιτόκια για όλους. Και δεύτερον, η δεύτερη γραμμή είναι να μειώσουμε το φορολογικό έλλειμμα κατά τρόπον ώστε να μειώσουμε ε, το, ε, το κόστος των ασφαλίστρων κινδύνου και των επιτοκίων. Επίσης δεν πρέπει να μειώσουμε, ε, ε, πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Και τώρα ο κύριος Ντομινίτσι. Καλημέρα κύριε Δικητά και σας καλωσορίζουμε στην αίθουσά μας. Απαντήσατε εν μέρη ε, στις ερωτήσεις ε, σχετικά ε, με τις οτιμίες ε, και με την ανταγωνιστικότητα. Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου κυρίου Τρισέ, η μόνη δυνατότητα έτσι ερμηνεύτηκε τουλάχιστον από, τις, ε, από τους οίκους αξιολόγηση να αυξηθούν τα επιτόκια και μόνο ο υπενιγμός αυτός προκάλεσε αλυστοιτές αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή ζούμε λοιπόν μια συγκεκριμένη κατάσταση και οι απαντήσεις ε, που δίνεται σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται και συναρτώνται από τον κίνδυνο αύξησης πληθωρισμού στις χώρες του Βορρά. Αυτό όμως θα είχε άμεσες επιπτώσεις ε, στις χώρες του αποκαλούμενου νότου της Ευρώπης. Είναι λοιπόν ε, σαφές ότι σαφώς ε, και δεν πρέπει κανείς να πειράξει τι συναλλαγματικέ ισοτιμίε. Όμως εγώ θεωρώ ότι η μείωση του χρέους δεν αρκεί για να προκαλέσει κανεί ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Αν λοιπόν υπάρχει επαγγελματική υπευθυνότητα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Δηλαδή ο κίνδυνος να επιμερίζεται, να μειωθεί γενικά το εξωτερικό χρέος, να υπάρχει μια πιο ουσιαστική πολιτική. Και η δική μου ερώτηση είναι εξής. Έχετε την αίσθηση ότι οι θεσμοί γίνονται σεβαστοί. Εσείς είπατε εξάλλου και σε γραπτή μορφή σε ερωτήσεις, που σας ετέθησαν ότι είσαστε dedicated European, αφοσιωμένος και στρατευμένος Ευρωπαίος. Ερωτώ λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν πράγματα και πέρα από το συνηθισμένο. Θεωρείτε λοιπόν ότι το καθήκον ενός ε, μελλοντικού Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, είναι να προβεί σε αυτές τις ε, ειδικέ ενέργειες πέρα από αυτά που είναι τα θεσμικά όρια για να μπορέσει ακριβώς να δρομολογήσει την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και στην αρχή, ε, τη δική μου τη ζωή σε μεγάλο βαθμό την αφιέρωσα στην οικοδόμηση της Νομισματικής Ένωσης και της Ευρώπης. Πάρα πολλά λοιπόν από τα προβλήματα τα οποία βιώνουμε σήμερα και νομίζω αυτό λίγο πολύ το γνωρίζουν όλοι, πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα ανάγονται στο γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Δηλαδή, ε, φτιάξαμε μια νομισματική ένωση, έχουμε το κοινό νόμισμα, πολλές χώρες ε, θεώρησαν ότι αυτό αρκεί. Μετά όμως ξαφνικά ανακάλυψαν ότι αυτό δεν αρκεί για να επιτύχουμε την νομισματική ένωση, δεν αρκεί αν δεν εφαρμόζονται και οι δέουσες πολιτικές. Η διαδικασία λοιπόν η πολιτική πρέπει να επανεξεταστεί, να μελετηθεί. Τώρα βρισκόμαστε στο μέσο του κυκλώμα, κυκλώνα. Κατά την άποψή μου, το αμέσως επόμενο βήμα είναι να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό που ήδη έχουμε. Ε, να το πω πιο ξεκάθαρα. Είχαμε ένα σύστημα ρυθμίσεων. Stability and Growth Pact το μηχανισμό σταθεροποίηση για την δημοσιονομική πειθαρχία. Πέντε χρόνια πριν αποδυναμώσαμε αυτόν τον οργανισμό, αυτόν τον μηχανισμό μάλλον, και αυτό ήταν λάθος. Πρέπει λοιπόν να επαναφέρουμε κανόνες ε, πειθαρχία και μιλώντας για πειθαρχία αναφέρομαι κυρίως σε προληπτικούς κανόνες εποπτείας και σε κυρώσεις. Κυρώσεις που θα είναι πολιτικές ε, αλλά και δημοσιονομικές έτσι ώστε να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία. Γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Προέδρου κ. Τρισέ και εγώ συμμερίζομαι απόλυτα αυτές ε, τις απόψεις. Να είναι αυτόματες οι διαδικασίες ακριβώς για να αποφύγουμε την εμπειρία που κάναμε με το σύμφωνο σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε πάρα πολύ και με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπόρεσε τελικά να ξεπεράσει τους προηγούμενους δύσκολους μήνες. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν η λέξη κλειδί όλης αυτής της διαδικασίας είναι ενίσχυση, εμβάθυνση, διεύρυνση. Ενίσχυση της εποπτείας, ε, όπως ακριβώς σας το περιέγραψα τώρα, εμβάθυνση με την έννοια να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες και διεύρυνση, η διαδικασία του ελέγχου και των ρυθμίσεων να επεκταθεί και σε άλλους τομείς που δεν είναι μόνο η δημοσιονομική πειθαρχία. Ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα πάρα πολλών κρατών σήμερα είναι η ανταγωνιστικότητα, η οποία αυξάνεται όμω με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Στον τομέα βέβαια των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέχρι ε, να υπάρξει πρόσφατα αυτή η συμφωνία που ήταν το αποτέλεσμα της ομάδας εργασίας του κ. Βαν Ρομπόη. Πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, εισαγάγαμε κοινού κανόνε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτοί οι κανόνε δεν είναι ακόμα δεσμευτικοί. Θα ήταν καλύτερα να σκεφτούμε να κάνουμε του κανόνε αυτού ε, δεσμευτικού, Με άλλα λόγια δηλαδή, να εφαρμόσουμε τα στοιχεία δημοσιονομικής πειθαρχίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και σε άλλους τομείς. Είναι λοιπόν αυτό, αυτή ε, είναι μια ρεαλιστική διαδικασία. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε ένα άλμα προς τα μπρος. Με νέους οργανισμούς, νέες απόψεις θα πρέπει να γνωρίζουμε την κατεύθυνση που ακολουθούμε. Όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τα βήματα εκείνα τα οποία ρεαλιστικά μπορούμε να ε, επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων ο κύριος Κλίντς. Mm. Κύριε Ντράγκη, την απάντηση στο πέμπτο ερώτημα είπατε ότι ε, θέλετε να έχετε κατευθυντήριες γραμμές για την ε, νομισματική σταθερότητα, για την ανεξαρτησία της ΕΚΤ και μιλήσατε στο 3 για μεγάλο πραγματισμό σχετικά με το οικονομικό περιβάλλον. Διαπιστώνουμε όμως ότι η ε, η ανεξαρτησία της ΕΚΤ ε, δεν υπάρχει πλέον κατόπιν της ε, ε, κρίσεως για να μπορέσει να αμυνθεί της σταθερότητος του νομισματικού τομέα και αυτό οφείλεται σε συμφωνίες και συμμαχίες που επετεύθηκαν με, την, με τον πολιτικό χώρο. Οπότε εάν μιλάμε συνέχεια για ανεξαρτησία de facto της ΕΚΤ και αν μιλάτε για healthy πράγμα της που λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές συνθήκες δεν νομίζετε ότι υπερβάλλεται. Ευχαριστώ. Κύριε Κλίντς. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια ο ρεαλισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την έννοια της στρατηγικής εξόδου δεν θα συμφωνήσω μαζί σας για το γεγονός ότι έχει απεμπολίσει την ανεξαρτησία της η ΕΚΤ, διότι η ΕΚΤ έχει αναλάβει μία σειρά μέτρων όπως το πρόγραμμα της αγοράς χρεογράφων και την χρηματοδότηση, την συνεχή χρηματοδότηση των τραπεζών, ένα σύστημα για το οποίο αλλάζουμε όνομα κάθε μέρα, δηλαδή ε, για τις τράπεζες που εξαρτώνται υπερβολικά από την ε, ε, κάλυψη της ρευστότητός τους από την ΕΚΤ. Και σε όλα αυτά βασιζόμαστε σε μία ουσιαστική ιδέα. Εάν δηλαδή τα μέτρα αυτά δεν είχαν αναλυφθεί ορισμένα ε, από τα δίκτυα επικοινωνίας της νομισματικής πολιτικής θα είχαν ε, νεκρωθεί και γι' αυτό πάντοτε ε, πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα νομισματικής πολιτικής. Αυτό είναι πολύ βασικό, διότι άπαξ ε, και ε, αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει πλέον ο, κίνδυνος αυτός, θα πρέπει να αλλάξουμε ίσως επίσης όσον αφορά το πρόγραμμα των αγορών χρεογράφων το άλλο πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε για όλα αυτά τα μέτρα ήταν ότι ήταν μέτρα που είχαν επινοηθεί σαν προσωρινά και κανένα δεν επρόκειτο να διατηρηθεί. Το τρίτο θέμα είναι ότι κανένα από αυτά τα μέτρα δεν αμφισβητεί τους στόχους μας του να εξασφαλίσουμε την μεσοπρόθεσμη ε, σταθερότητα των τιμών για όλη την Ευρωζώνη. Και η ΕΚΤ κατάφερε να ε, επιτύχει την ε, σταθερότητα των τιμών σε επίπεδο του 2% και χαμηλότερα κατά όλη την περίοδο της κρίσεως. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνούμε διότι στην εποχή αυτή του 2008, του 2009 και ενός μέρος του 2010 καταρτήσαμε ένα σύστημα το οποίο μπορούσε ε, να καθυλώσει ε, τις ε, προσμονές πληθωρισμού και επέτρεψε στην ΕΚΤ να διατυπώσει μια πολιτική εξόδου από την κρίση. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των τιμών και άρα η ΕΚΤ έχει παραμείνει ανεξάρτητη. Όπως όμως σωστά είπατε πρέπει να υπαγρυπνούμε και πρέπει να δούμε και να θυμόμαστε για ποιο λόγο αναλάβαμε αυτά τα μέτρα. Για να είμαι ακόμη πιο ομός. καμία κρίση κυρίαρχου χρέους ούτε ε, καμία τράπεζα η οποία θα επιμένει να ε, προβαίνει σε συναλλαγές δεν μπορεί ε, να εμποδίσει την έκτα από το να διατηρήσει την πολιτική της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δίκητά. Θέλω καταρχάς να σας ευχηθώ ότι το καλύτερο τους τραγμένους αυτούς καιρούς Πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι η ΕΚΤ έθεσε τον εαυτό της σε μια κατάσταση όπου ως ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα συναποφασίζει και συμπροετοιμάζει δημοσιονομικά μέτρα για να ληφθούν στην κυρίαρχη Ελλάδα, σε ένα κυρίαρχο κράτος όπως την Ελλάδα, όπως την ιδιωτικοποίηση ελληνικών περιουσιακών στοιχείων. Δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι επικίνδυνο για το μέλλον, ότι προδικάζει το μέλλον, ότι είναι επικίνδυνο προηγούμενο. Δεν μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της ΕΚΤ όταν αποτελεί αυτή πια τμήμα της πολιτικής λύσης του προβλήματος του ελληνικού χρέους. Θα συμφωνούσα μαζί σας ως προς το τελευταίο τμήμα, δηλαδή αν η ΕΚΤ γινόταν τμήμα της πολιτικής λύσης που απαιτείται, τότε αυτό θα την έκανε καθεαυτό να χάσει την ανεξαρτησία της, αλλά απλώς συμμετέχει σε διάφορα επεισόδια αντιμετώπισης της κρίσης με ρόλο αξιολόγησης των πιθανών κινδύνων και δημοσιονομικών αναδιαρθρώσεων καθώς και ρόλο επιτήρησης κυρίως δε αξιολόγησης της βιωσιμότητας των χρεών. Αυτό δεν διαφέρει πολύ από άλλες ανάλογες καταστάσεις, αλλά αν σήμαινε αυτό ότι και πολιτικά εμπλέκεται, τότε θα είχατε δίκιο. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να μην ξεπεράσουμε την εντολή μας και να μην μπούμε σε χωράφια άλλα από αυτά που έχει αναλάβει η επίσημος η Ευχαριστούμε. Και τώρα εξ ονόματος των Πρασίνων ο κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ Σάρων. Κύριε Ντράγκη, ίσως είστε ο πιο ορθόδοξος καθολικός που έχω ποτέ συναντήσει. Βλέπω από το βιογραφικό σας και τις δηλώσεις σας ότι θέλετε να παραμείνει ανεξάρτητη, ανεξάρτητη η ΕΚΤ. Αλλά και εγώ θα ήθελα να προασπιστώ της δικής μας ανεξαρτησίας ως νομοθετών που είναι υπόλογοι προς το λαό ενώ εσείς όχι. Είπατε να προσέξουμε να μην ξεπεράσουμε την εντολή μας. Η ΕΚΤ όμως το κάνει αυτό καθημερινά. Γιατί όταν λέει, όπως είπατε και εσείς σήμερα, ότι πρέπει να προστατέψουμε τους δημόσιους επενδυτές και πιστωτές και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα μεταφέρουμε το βάρος ή τον κίνδυνο του χρέους σε δημόσια χέρια κάνετε μια πολιτική επιλογή. Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί, αλλά είναι πολιτική επιλογή, δεν είναι τεχνική επιλογή. Όταν η ΕΚΤ διαστόματος Ζαν Κλοντ Τρισέ, δεν ξέρω αν θα κάνετε και εσείς το ίδιο, συνήθως έτσι γίνεται, ζητάει περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και αυξήσεις της φορολογίας και αυτό είναι πολιτική επιλογή η εξισορρόπηση των προπολογισμών είναι ένα πράγμα, αλλά μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και συνήθως η ΕΚΤ ζητάει τον α τρόπο αντί του β. Κάνει επιλογές δηλαδή. Επομένως, ούτως ή άλλως, είτε είναι μέλος είτε όχι της Τρόικας η ΕΚΤ, κάνετε πολιτικές συστάσεις και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Θα ήθελα και εγώ να περιοριστείτε στην εντολή σας που είναι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Πώς θα διασφαλίσετε λοιπόν ότι πράγματι δεν θα ξεπεράσει την εντολή της Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ. Τρία σημεία θίξατε. Πρώτον, είμαστε υπόλογοι στους πολίτες της Ευρώπης και σε εσά, στους ευρωβουλευτές. Γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ. Και γι' αυτό θέτετε το ερώτημά σας. Δεύτερον, δεν είπα ποτέ ότι θα προστατεύσω τους ιδιώτες επενδυτές. Όχι, όχι. Εσείς το θεωρείτε δεδομένο, αλλά εγώ δεν το είπα ποτέ. Εκτός αν το είπα ασυνείδητα που δεν πιστεύω. Υπάρχουν τρεις τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς το ελληνικό πρόβλημα. Η πτώχευση, η ανταλλαγή χρεών και το κούρεμα. Και αν υπάρξει credit default, τότε αυτό σημαίνει ορισμένες επιπτώσεις. Και θα ήθελα να τις ξέρετε τις επιπτώσεις μιας στάσης πληρωμών. Δεν το απαγορεύω, απλώς να ξέρετε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Εμένα καθήκον μου είναι να σας γνωστοποιήσω ποιες είναι οι επιπτώσεις. Τρίτον τώρα, για τη φορολογία και τις δαπάνες. Γιατί ενδιαφέρεται η ΕΚΤ για την ανάπτυξη. Γιατί ενδιαφέρεται για την ανταγωνιστικότητα. Ο λόγος είναι ότι ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλό χρέος η ανάπτυξη συμβαδίζει με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Είναι απαραίτητη για να υπάρξει σταθερότητα. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη δεν αποπληρώνει κανείς τα χρέη του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να υπάρξει ανάπτυξη λοιπόν χρειάζονται ορισμένα πράγματα και άλλα που πρέπει να αποφευχθούν. Μπορώ να σας τα αναφέρω με τη σειρά, αλλά αυτή είναι η λογική την οποία ακολουθούμε εμείς στην ΕΚΤ για πράγματα που σε πολλούς όπως και σε εσά φαίνονται ξένα προς τον τομέα με τον οποίο ασχολείται μια κεντρική τράπεζα. Είστε πολύ ορθόδοξος καθολικός φαίνεται. Τώρα το ΕΛΚ ο Αλφρέδος Παλώνε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Δικητά, ε, προηγουμένως μιλήσατε για τη σχέση που υπάρχει ε, στην κρίση που αντιμετωπίζει η Ιταλία ε, με την κρίση που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Η απάντησή σας με ικανοποίησε, όμως θέλω να πω το εξή. Η κατάσταση αντικειμενικά είναι τελείως διαφορετική, δηλαδή από αυτό που υπήρχε χθε με αυτό που υπάρχει σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε να κάνουμε με την παγκοσμιοποίηση, έχουμε να κάνουμε με την αλληλένδεση των αγορών, των οικονομιών, Άρα δηλαδή ε, βγαίνουμε από, μία, από τις χειρότερες κρίσεις ε, που υπήρξαν ποτέ. Και ε, σε αυτή την κρίση από αυτή την κρίση προέκυψε ότι υπάρχουν και όρια. Όρια των διεθνών ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Ε, υπάρχουν κερδοσκοπίες, ε, ασύστολες κερδοσκοπίες, πέρα λοιπόν από οποιοδήποτε, οποιαδήποτε δυνατότητα ελέγχου των κρατών. Βλέπουμε ότι όλα αυτά οδήγησαν στο να υπάρχει η ευαίσθητη αυτή κατάσταση σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο. Και ρωτώ το εξή, κύριε Δικητά, εσεί πώ πιστεύετε ότι πρέπει να χαράσετε η νομισματική πολιτική έτσι ώστε να μην βρίσκεται σε αντίφαση με την αναγκαιότητα πιθανότητα να υπάρχει ε, σταθερότητα των τιμών και χρηματοπιστωτική σταθερότητα κυρίως. Όταν ξέσπασε η κρίση, πάρα πολλοί είπαν ότι οι νομισματικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι το 2007 οι πολιτικές αυτές δεν έλαβαν επουδενή υπόψη τους ε, τις ε, κερδοσκοπικές ε, φούσκες, τις πομφόλιγες. Δεν έκαναν τίποτα για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Υπήρχε ένας μεγάλος κεντρικός τραπεζίτης στην Αμερική που έλεγε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν θα σπάσει η φούσκα, απλά θα απομακρύνουμε τα πτώματα. Άλλαξε όμως η κατάσταση. Τώρα πλέον κανείς ε, δεν θεωρεί ότι μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσε να είναι στρατηγική νομισματική. Γιατί επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, πρώτος στόχος νομισματικής πολιτικής είναι μεσοπρόθεσμα να σταθεροποιηθούν οι τιμές. Όμως θα πρέπει να έχει κατά νου και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Όπως ε, το βιώσαμε εξάλλου και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όμως ε, η νομισματική πολιτική αυτή καθεαυτή δεν είναι το καλύτερο μέσο για να αντιμετωπιστούν προβλήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικά εργαλεία, όπως παραδείγματος χάρη με το εργαλείο που αποκαλείται μακροπροληπτική ρύθμιση. Οι πολιτικές αυτές δεν είναι σε αντίφαση μεταξύ τους. Είναι δύο πολιτικές που συμπληρώνονται. Η νομισματική πολιτική που διασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών διασφαλίζει και τα το πίσω μέρος της ε, ε, ρύθμισης. Διότι όταν ξεφεύγει ο πληθωρισμός, αυτομάτως ε, δημιουργείται αστάθεια. Γι' αυτό λοιπόν η νομισματική πολιτική πρέπει να εκτελέσει, επιτελέσει το καθήκον της και κάνοντας αυτό θα πρέπει να έχει κατά νου και το ενδεχόμενο κάποιες επιτάχυνσεις που μπορεί να προκύψει σε κάποιους τομείς της οικονομίας. Όταν λοιπόν συζητάμε για νομισματική πολιτική πρέπει να έχουμε κατά νου παραδείγματος χάρη τι συμβαίνει στον τομέα των ακινήτων ε, ή στο ευρώ ή στις, ε, στα δάνεια που χορηγούνται ή να έχουμε κατά νου ε, κάποιες προϋποθέσεις. Λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά σε σχέση με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και με τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Όμως ο στόχος είναι διαφορετικός. Ο στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών. Και μαζί με αυτό υπάρχει και ένα άλλο εργαλείο που είναι το εργαλείο της μακροπροληπτικής ρύθμισης. Θα αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Σήμερα ας πούμε, αν δούμε ότι σε, έναν, σε ένα τμήμα της Ευρωζώνης διαμορφώνεται μία φούσκα ακινήτων, ένας τρόπος για να τα αντιμετωπίσει κανείς είναι να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 το κομμάτι εκείνο ενός ακινήτου που δεν χρηματοδοτείται από την τράπεζα, δηλαδή loan to value ratio ή αν θέλετε τα δάνεια των τραπεζών να είναι ανάλογα με το εισόδημα εκείνου που παίρνει το δάνειο. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα εργαλεία ή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί κανείς να αυξήσει το κεφάλαιο των τραπεζών. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ενός, ένα τελικό παράδειγμα πρόσφατο που προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας ε, εποπτείας διαπιστώθηκε ότι μια Ιταλική τράπεζα είχε επενδύσει πάρα πολύ στον τομέα των ακινήτων και η ρυθμιστική αρχή ζήτησε από αυτή την τράπεζα να αυξήσει το κεφάλαιό της. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα ε, πρόληψης, ε, ρύθμισης και μακροπροληπτικής ρύθμισης. Και θέλω να πω και μελαμβάνω δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις πολιτικές που σας προέγραψα, περιέγραψα προηγουμένως. Κύριε Ντράγκη, η κυρία Μακάρθη, με ενδιαφέρει η δικιά σας άποψη και όχι αυτή των προκατόχων σας στην ε, ΕΚΤ. Ξέρω ότι έχετε απορρίψει την ιδέα του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά είπατε ότι συμφωνείτε με τους στόχους. Δέχεστε λοιπόν ότι ο τομέας αυτός των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν φορολογείται παρκών και η ΕΚΤ ε, αυξάνει τη τις αμοιβέ ε, χωρίς να συμβάλλει εις, ε, τις, εις ε, την πραγματική οικονομία και θα ακούσετε τους πολίτες σας εφόσον είστε υπόλογος προς αυτούς και θα λάβετε η υπόψη σας το θέμα για την εφαρμογή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Επίσης στον τομέα αυτό θα επιζητήσετε να υπάρξει μια παγκόσμια συνένεση στην εφαρμογή του μέτρου αυτού. Σχετικά με ε, τον φόρο ε, χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών, επαναλαμβάνω αυτό που είπα, θέλουμε να καλύψουμε τους σωστούς στόχους του μέτρου αυτού. Θέλω να το διερευνήσω περισσότερο. Δηλαδή, με ένα παράδειγμα, πιστεύω ότι στο ΣΥΦΙΣ ε, οι συστημικές ε, οικονομικές, ε, τα συστημικά θεσμικά όργανα στον τομέα της χρηματοοικονομίας πρέπει να επιζητούν δύο στόχους. Καταρχάς, να μας αποτρέψουν από την που πήραν οι Lehman Brothers. Δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρξει μια χρεοκοπία τραπέζης η οποία θα πληρωθεί από τους φορολογούμενους και ο δεύτερος στόχος είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει μια τραπεζική χρεοκοπία η οποία να οδηγήσει σε μια διαταραχή σαν αυτή που δημιούργησε η Lehman. Αυτό ο, λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο έργο που αναφέρεται ακριβώς στη λειτουργία αυτών των θεσμικών οργάνων και βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Καταρχήν, τα θεσμικά αυτά όργανα πρέπει να έχουν δυνατότητα μεγαλύτερης απορρόφησης, δηλαδή να έχουν μεγαλύτερο αποθεματικό κεφαλαίου από, εφόσον είναι συστηματικά σημαντικά ε, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, διότι ε, είναι μεγάλες τράπεζες, μπορεί ε, να είναι συνδεδεμένες, να είναι αναντικατάσταση είναι μέρος του συστήματος. Χρειάζονται λοιπόν περισσότερο κεφάλαιο καλής ποιότητος κατά τρόπον ώστε να μπορούν όντως να απορροφήσουν τους κραδασμούς. Εάν α, χρεοκοπήσουν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ε, χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των φορολογουμένων. Θα υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα διαχείρισης κρίσεως που θα μπορέσει να διαχειριστεί την χρεοκοπία. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει πολλά πράγματα εκ των οποίων δύο είναι πολύ βασικά. Καταρχήν, ότι ε, αν αποτύχει μια πολύ και χρεοκοπήσει μια πολύ μεγάλη τράπεζα θα πρέπει να μπορέσουμε να γνωρίζουμε ποια τμήματα πρέπει να κλείσουν αμέσως σε αυτήν την τράπεζα και ποιοι τομείς πρέπει να διατηρηθούν ανοιχτοί και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ουσιαστικές λειτουργίες της τράπεζας πρέπει να παραμείνει ανοιχτό ε, δηλαδή οι καταθέσεις, οι ε, πληρωμές και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων έχοντας υπόψη ποιος τελικά θα χάσει χρήματα εάν θα ε, αποτύχει η τράπεζα διότι πρώτα θα είναι σε περίπτωση χρεοκοπίας τραπέζι θα χάσουν οι μέτοχοι και δεύτερον οι χρηματοδότες, δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πιστωτές, ποιοι είναι οι πιστωτές που θα πρέπει να προστατευτούν, οι καταθέτες θα πρέπει να προστατευτούν και μέχρι ποιο επίπεδου και ούτω καθεξής. Οι μεγάλοι ανασφάλιστοι πιστωτές επίσης θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι και το βασικό είναι ότι θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε και να εργαζόμαστε βάσει της ιδίας λίστας, διότι είμαστε μία ένωση θα πρέπει να συμφωνήσουμε συλλογικά και τρίτον είναι το θέμα της εποπτείας. Χρειάζεται μία πιο ανεξάρτητη και πιο ερευνητική εποπτεία από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και υπάρχουν πολλές προτάσεις επ' αυτού όσον αφορά την εντολή να έχουν περισσότερες εξουσίες οι επόπτες και ούτω καθεξής. Ε, αυτά καλύπτονται από το σύστημα ΣΥΦΗ και πρέπει να σας πω σε τι απευθύνεται ο φόρος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αφού ξεπεράσουμε τις δυσκολίες εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος, στο νέο σας ρόλο. Είσαστε έτοιμος να αναλάβετε όλες αυτές τις λειτουργίες και να αποφασίσετε διότι όλοι συμφωνούν ότι οι τράπεζες υποφορολογούνται αυτή τη στιγμή. Βεβαίως είμαι πρόθυμα, αλλά πρέπει να δω ποιες θα είναι οι εξωτερικές επιπτώσεις της εφαρμογής αυτής της φορολογίας. Είμαι έτοιμος να εξετάσω τις εναλλακτικές λύσεις μπορώ να συνεχίσω επί του θέματος αλλά ουσιαστικά εξετάζουμε αυτές ε, τις, ε, ε, τις λύσεις τώρα και αν έχετε κάτι να προτείνετε συγκεκριμένα θα κοιτάξουμε τις εναλλαγές. Τώρα όλε Σμίτ. Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Μέχρι τώρα Είμαι ε, φιλελεύθερος από τη Σουηδία, εκτός Ευρωζώνης. Μέχρι τώρα λοιπόν πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα από τις απαντήσεις σας. Στις γραπτές σας ε, απαντήσεις ε, σε σχέση με την ίση εκ περιτροπής ανάληψη προεδρίας στην ε, ΕΚΤΑ ανεξάρτητα από εθνικότητα ή φύλλο. Η απάντησή σας είναι ε, άμεση και ορθόδοξη θα έλεγα είπατε ότι κάτι τέτοιο ε, δεν είναι παραγωγικό δεν μπορεί έτσι κανείς να επιλέξει τον καλύτερο κατανοώ αυτό που λέτε κύριε Τράγκη παρότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ικανές γυναίκες και στον τομέα της νομισματικής πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν ε, ρωτώ, πιστεύετε ότι θα ήταν πρόβλημα για την ΕΚΤ να έχει ανοιχτό διάλογο με το κοινό και να ανακτήσει την ε, προσέγγιση στους πολίτες. Τη στιγμή όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν εφόσον δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι όλοι άντρες και δεν αμφισβητώ τις ικανότητές σας κύριε Ντράγκη, ε, που δεν είναι, αλλά ε, εδώ ίσως υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Και το λέω και εγώ ε, και μην ξεχνάτε ότι έρχομαι από μια άλλη χώρα. Ίσως εσείς ε, να είσαστε και μισός Γερμανός, αλλά είμαστε του ιδίου φίλου. Απάντηση του κυρίου Ντράγκη. Νομίζω έχετε δίκιο πράγματι. Υπάρχει πρόβλημα με την έννοια ότι... Το πρόβλημα αυτό είναι γενικότερο. Έχουμε όμως ε, μια συνθήκη, έχουμε μια εντολή η συνθήκη δεν λέει ότι πρέπει να προβλέπεται μία ποσόστοση ανάλογα με το φύλλο ή την ε, εθνοτική προέλευση. Ε, η συνθήκη λέει ότι ε, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή γενικότερα τα μέλη αυτής θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τα επαγγελματικά τους προσόντα. Αυτά λέει η συνθήκη. Βεβαίως ε, οι ηγέτες μας ε, ε, θα έπρεπε ίσως να έχουν αυτό το θέμα που θίξατε κατά νου για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και γενικότερα συμφωνώ και επαυξάνω με αυτά τα οποία είπατε. Και για μένα είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι πρόβλημα για όλους που έχουν συνειδητοποιήσει κατά κάποιον τρόπο το πρόβλημα και αναμφισβήτητα αυτό αποτελεί πρόβλημα για μένα. Το ότι δεν υπάρχουν γυναίκες. Πάντως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Banca d'Italia, της Κεντρικής Τράπεζας Τελεία, ε, να σας πω ότι υπάρχει μία γυναίκα. Μόνο μία, λέει η πρόεδρος. Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα θα προχωρήσω στο ε, ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υποψήφιε. Θα προσπαθήσω να ε, βασιστώ εις την ε, την βάση και θα ξεκινήσω από την αρχή σημαίνει ότι ε, θα πρέπει κατά 16,5% για την Ελλάδα να μειωθούν τα δημόσια έξοδα τα δημοσιονομικά έξοδα και αυτό συνδυάζεται με ανεπαρκή ε, ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι ε, δεν είστε υπέρ της αναδιάρθρωσης. Και ε, σήμερα ε, μία διάσωση έχει επικυρωθεί και ίσως όμως χρειαστεί άλλη μία μετά από λίγο καιρό και ορισμένα κράτη-μέρη δεν είναι υπέρ του να υπάρξει μία τέτοια διαδικασία η οποία μπορεί να διευκολύνει ε, την ε, αναδιάρθρωση. Αναρωτιέμαι λοιπόν ε, για αυτά που ελέγχθησαν γιατί δεν είναι δυνατό να υπάρξει αναδιάρθρωση και τι θα γίνει για να αντεπεξέλθουμε από αυτό το αδιέξοδο. Η ερώτηση είναι ότι ε, αυτοί οι οποίοι επεμβαίνουν στο Λουξεμβούργο ή αλλού επεμβαίνουν εις ε, το δεύτερο γενές επίπεδο του χρέους και ο Επίτροπος Ρεν είπε ότι τα κράτη δεν συμφωνούν. Ποια είναι τα τεχνικά προβλήματα και διαφορετικά τι είναι οι άλλες δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν διότι σε μερικούς μήνες θα επανέλθουμε στην κατάσταση αυτή η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει. Και πάλι αντιμετωπίζουμε περισσότερο το θέμα της χρηματοδότησης. Διότι ε, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε για να επιλύει προσωρινά προβλήματα και όχι για να υπάρξει μία φορολογική μεταφορά μεταξύ χωρών. Μπορεί ε, να αγοράσει ομόλογα ή ε, την ε, κύρια αγορά αλλά όχι στην δευτερεύουσα αγορά τα κράτη ενδεχομένως θέλουν να περιορίσουν τις δυνατότητες του μηχανισμού αυτού να μπορεί να επεμβαίνει στις αγορές ενδεχομένως και ε, να εμποδίσουν να συσσωρευτεί μεγάλο χρέος που έχει αγοραστεί στη δευτερεύουσα αγορά ε, χωρίς ε, αυστηρούς όρους όπως ισχύει στην περίπτωσή μας για να μπορέσει να είναι βιώσιμο το χρέος και είναι δυνατόν ένα τέτοιο σύστημα να λειτουργήσει στην, βασική, στην πρωτογενή αγορά διότι εάν θέλουμε ε, να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό σύστημα πρέπει εγώ να εξετάσω τι θα γίνει αν αρνηθούμε μια τέτοια λύση. Εάν υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να προβεί σε αγοραπολισίες στην δευτερογενή αγορά δηλαδή σε, ε, με επικουρικό τρόπο το ερώτημα είναι ότι πώς θα ελέγξω την αιρεσία των αγορών ή στη δευτερεύουσα αυτή αγορά. Μπορεί το ίδιο να συμβεί σε την κυρία αγορά. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς θα γίνουν αυτές οι συναλλαγές επί καθημερινής βάσεως ε, για λόγους πρακτικούς και όχι ίσως ε, ε, διανοητικούς. Κατά πολύ μεγάλο μέτρο λοιπόν θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Και τώρα ο Σάβιν Κούτας για την... Ε, Σας καλωσορίζουμε κύριε Ντράγκη. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων είναι η αρχή μιας μακράς σειράς ε, επισκέψεων, αλλά ας επανέλθουμε στα θέματα ανάπτυξης ε, στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι εμείς ε, ως σοσιαλιστές υποστηρίζουμε την ιδέα ένα τμήμα του δημόσιου χρέους να μετατραπεί σε ευρωομόλογα. Και επίσης ε, είμαι σίγουρος θα έχετε ακούσει για τα περίφημα project bonds όπως λέγονται. Και θέλω λοιπόν να γνωρίζω το εξής. Ε, ποια είναι η άποψή σας ε, ε, όσον αφορά στο να δημιουργηθούν ευρωμόλογα για να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη. Αυτό περίπου που έκαναν οι Ηνωμένε Πολιτείε για να χρηματοδοτήσουν το New Deal. Και ποια είναι η άποψή σα να χρησιμοποιηθούν ε, ομόλογα να εκδοθούν ομόλογα ανταλλάσσοντάς τα με απαιτήσει ε, χρέους. Αυτή την ερώτηση ήθελα να κάνω. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά ιδιομολόγων τα ε, growth bonds ε, είναι ομόλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την έννοια αυτή στηρίζονται από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, ως έχει η κατάσταση, βρισκόμαστε στα μέσα του ποταμού. Δεν έχουμε διασχίσει το ποτάμι για να πάμε σε μεγαλύτερη και πιο βαθιά ένωση. το θέμα λοιπόν ε, των κρατικών ομολόγων ή ενωσιακών ομολόγων, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι χώρες που έχουν πολύ καλή πιστοληπτική ικανότητα θα πληρώσουν περισσότερο και αυτές που έχουν κακή τελικά θα πληρώσουν λιγότερο. Έτσι λοιπόν, κατά κάποιον τρόπο, υπάρχει μια ανταλλαγή ανάμεσα στις χώρες και εδώ πρέπει να ελέγξει κανείς ότι κάτι τέτοιο είναι πράγματι συμβατό με την ρήτρα μη διάσωσης που υπάρχει στην συμφωνία. Παρεπιπτόντως, ε, το 1993 έγινε το λόγος για ομόλογα υποδομή infrastructure bonds. Αυτά τα είχε προτείνει τότε ο κύριος Ντελόρ και το θυμάμαι γιατί εγώ τότε ήμουνα σε αυτό το Συμβούλιο Κοφίν ε, που πρότεινε αυτά τα ομόλογα υποδομή. Και αυτά προκάλεσαν ε, βίε αντιδράσεις ε, πολλών κρατών και για τους λόγους που αντιμετωπίζουμε σήμερα μετά από 15-18 χρόνια, δηλαδή ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια ένωση όπου μεταφέρονται τα χρέη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ο κίνδυνο υπήρχε και ακριβώς πριν από 18 χρόνια. Για μένα λοιπόν ένα ευρωομόλογο είναι ένα απόλυτα νόμιμο εργαλείο. Μπορούμε να το σκεφτούμε αν θέλουμε να έχουμε μια ε, πιο συμπαγή ένωση. Μερικοί μίλησαν για ε, μίνι δημοσιονομική ένωση, αλλά δεν είναι αυτό, είναι κάτι παραπάνω. Εγώ λοιπόν σε αυτό Δεν ξέρω αν μου επιτρέπει ο κ. Λαμπέρ να το πράξω, αλλά θα ήθελα να τολμήσω να μπω σε πολιτικά χωράφια. Και θέλω να πω το εξή. Είμαστε μία ένωση. Άρα δηλαδή είτε μας δεσμεύουν κοινοί κανόνες, είτε είμαστε ενωμένοι από θεσμούς και από έναν προπολογισμό. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε τίποτα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είμαστε στην διαδικασία του να δεσμευόμεθα από κανόνες. Πρέπει να ενισχυθούν, να εμβαθυνθούν, να διευρυθούν οι κανονισμοί μας και όσο τα προσεγγίζουμε ο ένας τον άλλον, αυτές οι έννοιες θα αποκτήσουν και μεγαλύτερο βάρος. Εγώ ε, δεν ε, το βλέπω αντίστροφα, δηλαδή να υπάρχουν ομόλογα για να επιβάλλουμε την Δημοσιονομική Ένωση. Και βλέπετε εδώ ποιε είναι οι διαφορές στην πολιτική. Αυτό λοιπόν είχα να πω σε σχέση με τα τα Brady Bonds, αυτό είναι διαφορετικό, είναι ένα ε, χρηματοδοτικό εργαλείο για να αντιμετωπιστεί η δημοσιονομική κρίση και βασίζονται, όπως σας είπα, στην θελούσια ανταλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τοποθετηθεί ε, στο θέμα του πιστοτικού γεγονότος αν είναι ετελούς η ανταλλαγή δεν υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι στους οποίους αναφερθήκαμε και είπα όμως και προηγουμένως ότι κατά κάποιον τρόπο έχουμε μάθει ε, να αντιμετωπίζουμε λιγάκι τους κινδύνους. Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει κατά κάποιο τρόπο και τώρα εν ονόματι του ΕΛΚ η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτηση που ήθελα να υποβάλω στον κύριο Διοικητή είναι ακριβώς η ερώτηση που υπέβαλε ο προηγουμένος ο συνάδελφος. Σας ευχαριστώ και εγώ λοιπόν για την απάντηση αυτή που δώσατε. Με την ευκαιρία σας ε, κάνω ένα άλλο ερώτημα που έχει σχέση με την πρόταση ε, από τον κύριο Τρισέ ε, εκφράστηκε αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται για το, έναν Υπουργό Οικονομικών στην ε, Ευρωζώνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα θα έλεγα. Ε, είπατε ότι είμαστε σε μια διαδικασία που δεν είναι ολοκληρωμένη, χρειάζεται βάνθηση, συντονισμός, πάρα και από συντονισμό κεντρική πολιτική έχουμε ανάγκη βλέπουμε ότι και τα προγράμματα διάσωσης στις χώρες ε, που εφαρμόζονται παράδειγμα από τη δική μου χώρα δεν επιτυγχάνουν τους στόχους της ε, εργαλεία και πολιτικές παραπάνω χρειαζόμαστε. πιστεύετε ότι ένας υπουργός οικονομικών θα μπορούσε να δώσει μια προστιθεμένη αξία με όλες τις θεσμικές πέρα από τις πολιτικές δυσκολίες που μπορεί να έχει η δημιουργία αυτού του θεσμού αλλά πιστεύετε ότι θα μπορούσε να το δούμε θετικά βλέπαμε με δυσκολία την οικονομική διακυβέρνηση λίγα χρόνια πριν. Σήμερα είμαστε στο στάδιο της υλοποίησής της. Τι θα λέγατε για ένα βήμα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δεν έχουμε ακόμη οικονομική διακυβέρνηση. Κοντεύουμε, είμαστε στο σωστό δρόμο. όπως λέγαμε και πριν, πρέπει να ενδυναμώσουμε τους κανόνες μας, να τους ενισχύσουμε και να δεσμευτούμε περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα στους τομείς της δημοσιονομικής πειθαρχία, αλλά και της ανάπτυξης και των δομικών αλλαγών. Όπως για τα ευρωομόλογα πρέπει να προχωρήσουμε βήμα με το βήμα και μακροπρόθεσμα ό,τι και να σημαίνει αυτή η λέξη, πρέπει να υπάρξει ισχυρότερη κεντρική διακυβέρνηση πριν μπορέσουμε να σκεφτούμε το επόμενο βήμα. Πρέπει να καθησυχαστούν οι χώρες ότι εδώ δεν είναι ένωση μεταφορών. Και αυτό δεν θα διασφαλιστεί παρά αν υπάρξουν σοβαροί και αυστηροί κανόνες που δεν μπορούν να, να τυχαίνουν εξαιρέσεων. Ή τουλάχιστον όχι εύκολα οτιδήποτε επιφέρει αυστηρότερη επιτήρηση, αυστηρότερες κυρώσεις και αυστηρότερους κανόνες, σωστό θα είναι. Αλλά δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι για αυτό το θεσμικό βήμα όπως ένα ενωσιακό ομόλογο ή έναν αρμόδιο υπουργό εσωτερικά. Στο μέλλον όμως μπορεί. Ωραία. Τώρα για τους σοσιαλιστές η κυρία Περβάνς Μπερέζ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Διοικητά, και υποψήφιε μάλλον. Ίσως με θεωρήσετε παλαιομοδίτησα, αλλά εγώ θεωρώ ότι οι τράπεζες έχουν ως ρόλο τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Από το παρελθόν και την εμπειρία σας, που όλοι επενούν, μπορέσατε να ελέγξετε πολλές αγορές, αν και εξυπηρετούσατε και μία επιχειρήση των Goldman Sachs που δεν ανταποκρίνεται σε αυτόν τον στόχο. Η επενδυτική αυτή τράπεζα μέσω αυτορυθμίσεων ή απορυθμίσεων ε, κατάφερε να ελέγξει υπερβολικά την οικονομία χωρίς και μεγάλη διαφάνεια και με τα credit default swaps και τους διευθυντές της που έπαιρναν τεράστια πριμ ακόμη και ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε ότι πρόκειτο για αμοιβέ ε, όχι μεν παράνομες αλλά όχι και πολύ σωστές ε, αδίστακτες αμοιβέ. Εσείς θα μπορούσατε να λάβετε υπόψη σας την εμπειρία αυτή από τέτοιου είδους τράπεζες που στρέφουν τα νότα τους στην ενωσιακή πολιτική, στην πολιτική που χρειάζεται σήμερα η Ευρωζώνη. Όταν ήσασταν πρόεδρος του Φόρουμ για τη Σταθερότητα και του ESBF τον Μάρτιο την Άνοιξη γενικά του 2008 είχατε ζητήσει οι τράπεζες να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους απολογισμούς τους. Τι απολογισμό λοιπόν κάνετε τώρα ως προς αυτό. Οι τράπεζες ακολούθησαν τη σύστασή σας. Τέλος, σήμερα ως υποψήφιος μας μιλάτε αλλά δεν δέχεστε αυτά που είπε μία βραδινή εφημερίδα στη Γαλλία που έλεγε ότι είστε αντιπρόεδρος της Ευρώπης ε, για τη διαχείριση κυριάρχων κρατών. Τον δέχεστε αυτόν τον τίτλο ενώ η πρόεδρος Περβάνς παρακαλώ να τελειώνετε ενώ ένα αγγλικό περιοδικό δήλωσε ότι θα παρέμβεται ως κεντρική τράπεζα de facto σε κυβερνητική πολιτική. Λοιπόν, έχω δυόμιση λεπτά, οπότε ε, ήδη απάντησα για την εμπειρία μου στην Goldman Sachs. Εσείς μου λέγετε μου λέτε ε, όσο μπήκα στην Goldman Sachs. Ε, ίσως ξέρετε ότι σύμφωνα με το ανακοινωθέν τύπου ζήτησα να μην έχω επαφές με τις κυβερνήσεις λόγω του παρελθόντων μου και ήθελα μία περίοδο διακοπής μεταξύ της μιας δουλειάς στην άλλη. Το ερώτημα μου είναι εσείς αφισβητείτε το πρότυπο εργασίας του Goldman Μα, απαντάει ο κύριο Γκραγή, ε, έχουν 23.000 υπαλλήλου. Τι εννοείται business model. Πρέπει κανείς να παρακολουθεί αν ε, κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Κάποιο σχόλιο χωρίς μικρόφωνο με ρωτάτε για την, συνέντε, την ανακοίνωση που απάντησα και ουσιαστικά το ερώτημα αυτό έχει ήδη τεθεί και ξαναλέω ότι ήμουν, λειτουργήσα με ακαιρεότητα όσο εργαζόμουν στον Goldman Sachs και στο FSB ε, που υπήρξε μεγαλύτερη διαφάνεια το 2008. Κάναμε πολλή δουλειά και σήμερα ε, ο χώρος των ε, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διαφέρει πολύ από το 2006 με 8 αλλά τώρα πρέπει να εφαρμόσουμε τη Βασιλεία 3. Πρέπει να ε, δούμε πόσο θα εφαρμοστεί το σύστημα των τραπεζών, τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, θέματα που είναι ακόμη εν εξελίξη. Ο χώρος διαφέρει πάρα πολύ. Θα αποφύγουμε την επόμενη κρίση, δεν ξέρω, διότι έχουμε καταρτήσει κανόνες και συμπεριφορές που θα μας ενισχύσουν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στο μέλλον. Ε, με συγχωρείτε, αλλά μιλούν η πρόεδρος και ο υπερβός Περές συγχρόνως. Η πρόεδρος λέει, ε, ξεπέρασε στο χρόνο σου περβός και το λόγο έχει τώρα η κυρία Άστριντ Λούλινγκ. Ευχαριστώ κυρία πρόεδρε κατόπιν της παρατήρησης του συναδέλφου μου από τους φιλελευθέρους όλες Σμιτ για την ισότητα των φίλων θέλω να πω στον κύριο Ντράγκη ότι είμαι υπέρ της ισότητας των φίλων και προτιμώ μία γυναίκα η οποία είναι ικανή από έναν ανίκανο άντρα και αντιστρόφος. αλλά κύριε Ντράγκη δεν πρέπει να ντρέπεστε που είσαστε εμφανώς άνδρας όπως και όλοι οι επικεφαλής της ΕΚΤ. Θα ήθελα όμως ορισμένες διευκρινήσεις σε ορισμένα θέματα που θίξατε. Η ΕΚΤ αρνείται οποιαδήποτε αναδιάρθρωση η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ε, σαν ε, ένα πιστοτικό γεγονός ε, από τις αγορές. Αυτή η θέση οφείλεται στο ότι η ΕΚΤ η ίδια κατέχει δεκάδες εκατομμυρίων ελληνικών χρεογράφων δημοσιογράφων ε, και θα ήθελα να ξέρω αν αυτό επηρεάζει τη στάση της. Επίσης, όταν εάν ε, ε, τοποθετηθείτε στην ΕΚΤ σαν πρόεδρος θα τεθείτε στην ίδια θέση με τον κύριο Τρισέ και θα αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επιτροπή, επιστροφή εις της θέσεις ε, των κυβερνήσεων. Έχετε σκεφτεί δηλαδή ποια θα είναι η τακτική σας για να αντιμετωπίσετε τις εθνικές κυβερνήσεις. Βλέπω ότι επανερχόμαστε στο ερώτημα κλειδί της ημέρας αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέμα γιατί η ΕΚΤ στο έργο της έχει αυξήσει το πόσο είναι εκτεθειμένη προς την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και άλλες χώρες. Όταν λοιπόν η ΕΚΤ αποφασίζει και ε, παίρνει εγγυήσεις, οι εγγυήσεις αυτές κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες κινδύνου. Και μετά τα κουρέματα τα οποία εφαρμόζονται σε τέτοιες εγγυήσεις μειώνεται η αξία της εγγύησης ε, σε σχέση με τη στιγμή που προσεφέρθησαν σαν εγγύηση στην ΕΚΤ. Τα κουρέματα ε, προέρχονται από ε, κρίσεις στην τιμή αγοράς ή με τρόπο πολύ προσεκτικό. Αυτή τη στιγμή Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που αξιολογούν αυτά τα κουρέματα και οι θεσμοί αυτοί έχουν κοινούς κανόνες χρειάζεται δηλαδή μια πλατφόρμα για να υπάρξει μια τέτοια κίνηση και σας το λέω διότι τα εχέγγυα τα οποία έχουμε ήδη έχουν υποτιμηθεί και ε, Επίσης απορρίψαμε μία διεύρυνση των εγγύσεων αυτών στο τέλος του 2010 και θέλουμε να διατηρήσουμε τα ομόλογα αυτά μέχρι το τέλος της προθεσμίας τους και αν δεν υπάρξει μία κρίση στην αγορά δεν θα επηρεαστούν οι τιμές τους και οι αξίες τους. Υπάρχουν δηλαδή πολλές συλλογικές εθνικές ε, κινήσεις αλλά και οι εθνικές τράπεζες και η ΕΚΤ όλοι ε, προσέχουν διότι οι εθνικές τράπεζες θα πρέπει να, και αυτές να συμβάλλουν στο κόστος ε, ενός πιστοτικού γεγονότος σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στο σύνολο και αν δεν υπάρξει τέτοιο γεγονός ξέρουμε πού βρισκόμαστε όπως είπα και προηγουμένως. Αν υπάρξει ένα τέτοιο πιστοτικό γεγονός, ένα credit event, τότε όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αναδιόρθρωση ε, δεν θα είναι χωρίς συνέπειες για την επόμενη περίοδο. Διότι η ερώτηση που έθεσα στην αρχή των ερωταπαντήσεων που μου ετέθησαν ήταν ότι η Ελλάδα ε, θα έχει ε, ένα ένα έλλειμμα πέραν του 3% θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Εάν λοιπόν η στάση πληρωμών είναι επιλεκτική ε, και μη εθελοντική θα πρέπει να γνωρίζουμε το κόστος εάν επιλέξουμε αυτή την οδό. Και το τελικό ερώτημα... Από το ΕΛΚ, ο Γκέι Μίτσελ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τράγκη. Εσείς ε, συμφωνείτε ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται μια επιτυχία. Συμφωνείτε επίσης ε, ότι αυτή τη στιγμή η καλύτερη περίπτωση ε, για να υπάρξει επιτυχία είναι η Ιρλανδία η Ιρλανδική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο έχουν λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν το θέμα της ρευστότητας. Εσείς ε, περίπου 150 με 160 δις ε, θα ε, δανείσετε στην Ιρλανδία με απόδοση κάθε 14 ημέρες. Ένα πράγμα λοιπόν που μπορείτε να κάνετε για να επαναφέρετε την εμπιστοσύνη όχι μόνο στην Ιρλανδία αλλά στο σύνολο της Ευρωζώνης είναι ε, τα χρήματα αυτά ε, να γίνουν ε, η επιστροφή τους μακροπρόθεσμη, όχι ανά 14 ημέρες. συμφωνεί ότι κάτι τέτοιο είναι σωστό και θα έπρεπε να το εξετάσετε. Κοιτάξτε, ε, πρώτα απ' όλα πρέπει κανείς να πει το εξής, ότι στην Ιρλανδία από τότε που ξέσπασε η κρίση έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Ε, αν δεν κάνω λάθος, η Ιρλανδία είχε έλλειμμα ε, ισοζυγίου ε, τρεχουσών συναλλαγών της τάξης του περίπου 10% και τώρα έχει πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δηλαδή είναι ένα δείγμα ότι γίνονται πάρα πολλά. Τώρα, το θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι το εξής. Κατά πόσον το να χορηγήσουμε ένα εργαλείο, αν θέλετε, μεσοπρόθεσμο, κατά πόσον με τον τρόπο αυτό εισάγουμε ένα επιλεκτικό μέτρο πολιτικής το οποίο ενδεχομένως να είναι σε αντίφαση με το στόχο μας που είναι η σταθερότητα των τιμών. Δηλαδή, αν έχουμε μια, ένα εργαλείο μεσοπρόθεσμο, αυτό κατ' σημαίνει ότι χορηγούμε ρευστότητα σε μόνιμη βάση ανεξάρτητα από πληθωρισμό, ε, από προβλέψεις πληθωρισμού. Το λέω αυτό διότι αυτή είναι η βασική σκέψη που πρέπει να έχουμε κατά νου κάνοντας τις αξιολογήσεις μας που βεβαίω αν το κάναμε αυτό θα προσέφερε μια ασφάλεια στην Ιρλανδία υπάρχει και η άποψη ότι θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιούμε την νομισματική πολιτική για να επιβάλλουμε σταθερότητα τιμών. Το θέμα είναι ότι αν το κάνουμε βέβαια αυτό για μια χώρα, γιατί να μην το κάνουμε και για άλλες που βρίσκονται στην ε, περίπου ίδια κατάσταση. Και αν το κάνουμε για όλες τις χώρες, τότε πλέον δεν υπάρχει νομισματική πολιτική, τότε πλέον κολλάει η ρευστότητά μας και προσδιορίζεται σε μεσοπρόθεσμη βάση. Βεβαίω και γνωρίζουμε ότι αυτό θα αποτελούσε μεγάλη βελτίωση. Μην με παρεξηγείτε, απλά είμαστε αναγκασμένοι να σταθμίζουμε διαφορετικά ε, τα θέματα. Πολύ ωραία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ε, το κομμάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τώρα ε, πάμε στο επόμενο, το ESRB, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου. Ε, επειδή έχουμε τώρα κάποιο, κάποια πίεση χρόνου, θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις, θα τις οματοποιήσουμε και λέμε το ΕΛΚ, οι Σοσιαλδημοκράτες και οι ΆΛΔΕ να κάνουν μια ερώτηση και μετά να δώσετε την απάντηση. Ούντο, εσύ, εκ μέρου ε, των Σοσιαλδημοκρατών, γιατί δεν υπάρχει εδώ εκπρόσωπο ε, ε, του ΕΛΚ, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σα κάνω την ερώτηση στα γερμανικά. Να σα δώσω λοιπόν λίγο χρόνο για να μπορέσετε να ακούσετε την ερώτηση. Κύριε Ντράγκη, αυτή η Επιτροπή και αυτό το Κοινοβούλιο κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να ενισχύσουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κυρίως όσον αφορά στα καθήκοντα του Προέδρου σε σχέση με το Συμβούλιο Κινδύνων. Αυτή ήταν μια καλή επένδυση. Αυτό το δείξει βέβαια το μέλλον κατά πόσον ήταν σωστό αυτό το να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και θα σας εξηγήσω γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα λέω για τον εξή λόγο. Οποτεδήποτε εμεί επισημάναμε κινδύνους που απορρέουν από οικονομικούς παράγοντες, οποτεδήποτε το κάνουμε αυτό, τότε μας επενούν τα κράτη-μέλη αλλά και άλλοι για το ότι δείχνουμε ιδιαίτερη στράτευση, αλλά τελικά... Ε, μας λένε ότι επισημαίνουμε και στυλιτεύουμε λάθος φορείς και λάθος οργανώσεις. Όταν ας πούμε μιλάμε για τους οίκους αξιολόγησης, λάθος μας λένε. Ή όταν μιλάμε για τη βιομηχανία, πάλι μας λένε λάθος κάνετε. Όταν ε, οι συνάδελφοι κάνουν, ε, προβαίνουν σε πράξεις για το σορτάρισμα, για τα παράγωγα, πάλι μας λένε λάθος κάνετε. Ο συνάδελφος Λάμπερτ έχει δίκιο που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπερβαίνει συνεχώς τις αρμοδιότητές της ε, οποτεδήποτε προσαρμόζεται σε δημοσιονομικές ρυθμίσεις. Εμείς λοιπόν σας καλούμε στο μέλλον να διαδραματίσετε ένα διαφορετικό ρόλο, δηλαδή να ξεκινήσετε μαζί μας τον διάλογο για να βρούμε μαζί τα κρίσιμα θέματα. Και αυτή είναι η ερώτησή μου και η παρατήρησή μου επιτέλους βοηθήστε μας να σπάσουμε αυτό το ταμπού το οποίο ξεκινάει και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δήθεν εμείς όταν μιλάμε για τους κινδύνους που υπάρχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι πάντα επισημαίνουμε λάθος αίτια και λάθος φορείς. Ε, βοηθήστε μας να πούμε και κάτι σωστό, βοηθήστε μας να ξεφύγουμε από τη δίθεν αυτή επισήμανση λάθος φορέων. Πρόεδρος, ε, θα ομαδοποιήσουμε όπως σας είπα τις ερωτήσεις και μετά θα δοθούν οι απαντήσεις. Η Σιλβί. Ευχαριστώ. Όπως το είπε ο Ιντοπούλμαν, ε, πέρυσι παλέψαμε εδώ κατά τρόπον ώστε να υπάρξει ευρωπαϊκή εποπτεία κατόπιν της εκτίσεως Ντολαροζιέρ και τη εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό έχετε μισή ώρα παραπάνω εδώ διότι ε, σαν πρόεδρος ζητήσαμε να είστε επικεφαλής σαν πρόεδρος ΣΕΚΤ ζητήσαμε να είστε επικεφαλής της ομάδος ε, επιτήρησης του συστημικού κινδύνου και ε, με μία έκθεση η οποία χειροκροτήθηκε ευρέω, βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη κινήσεις κατά αυτής της ευρωπαϊκής εποπτείας. Μπορείτε σήμερα να δεσμευτείτε ότι θα υπεραμεινθείτε των προόδων που επιτύχαμε για να υπάρχει όντως ευρωπαϊκή εποπτεία διότι η έκταν είπατε έχει το προσωπικό, έχει την πείρα αλλά θα πρέπει να υπάρχει και το κύρος του Προέδρου της ε, σαν ε, Προέδρου ενός υπερεθνικού οργανισμού ε, επί ατόμων που ζητούν maximum organization με minimum requirements, δηλαδή όχι πολλά. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να δεσμευτείτε σήμερα ότι δεν θα υπάρχει οπισθοδρόμηση σχετικά με την ε, εποπτεία στην Ευρώπη και ε, ότι θα υπάρξει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και μέτρα και σταθμά ενιαία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Ευχαριστώ για αυτά που είπατε για τον έλεγχο των ανισορροπιών και πόσο σημαντικό είναι για τις χώρες να έχουν και άλλες δυνατότητες πέραν των χρηματοοικονομικών. Αναφερθήκατε στη Βασιλεία 3 που είναι το, κάτι που σας απασχολεί πολύ. Σχετικά με τη Βασιλεία την συνθήκη της Βασιλείας ε, και αναφέρομαι εις το ενιαίο σύστημα κανόνων και ότι ε, χρειαζόμαστε εθνικές εξαιρέσεις όταν στρεβλώνουν τη διαιτησία και πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, την σταθερό, χρηματοοικονομική σταθερότητα. Βλέπω λοιπόν όταν διαβάζω αυτό το έγγραφο ότι είναι αμφίσιμο. Είναι ένας πραγματικός εφιάλτης γιατί ε, από τη μία πλευρά ε, τονίζονται οι εθνικές τρευλώσεις, μειώνονται οι επιπτώσεις της θήκης της Βασιλείας και ε, η ανώτατη εναρμόνιση ζητείται σε ένα επίπεδο όπου τα κράτη δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά για να εξασφαλίσουν την χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Όταν λοιπόν μιλά κανείς για τους τραπεζίτες, μιλά στους τραπεζίτες και στους ηθήνοντες για τη Βασιλεία 3 μπορείτε να πρεσβεύετε τα ίδια επιχειρήματα εδώ και εκεί θα υπάρχουν απαντήσεις στο πρώτο σύνολο των ερωτήσεων και μετά θα επανέλθουμε. Καταρχήν στον κύριο Μπούλμαν δεν μπορώ να παρά να συμφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχει επικερδής διάλογος. Αυτή θα είναι η πηγή έμπνευσης για να ξεπεράσουμε αυτή την ε, ε, δύσκολη περίοδο για το, την εντολή της ΕΚΤ, για τον πολιτικό κόσμο και συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε συνείδηση του τι είναι η εντολή που έχουμε αναλάβει και να προσιλωθούμε σε αυτό. Δηλαδή να υπάρχει ένας επικερδής, επικοδομητικός και συνεχής διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προς την κυρία Γκουλάρ έχω να πω τα εξής. Ο συμβιβασμός Ντελαροζιέρ ήταν όντως καλός. Και οι περισσότεροι από μας θα ήθελαν κάτι το πιο φιλόδοξο ίσως αλλά τελικά αυτό ήταν εφικτό και θα αναθεωρηθεί κατά καιρού. Οπότε πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί. Πρέπει να δούμε εάν οι εξουσίες τις, ε, οι οποίες θα ανατεθούν στα διάφορα όργανα είναι επαρκή διότι οι πόροι θα αυξηθούν ιδιαίτερο για τον μηχανισμό παρέμβασης αλλά βεβαίως εάν ε, δεν συνεργαστούμε με τους εθνικούς επόπτες όποια συστήματα και να καταρτήσουμε δεν θα λειτουργήσει ποτέ το σύστημα και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι καταρχήν να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να υπάρχει μία αξιολόγηση από τους ομολόγους ε, μεν των δε, να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει αξιοπιστία και πιστεύω ότι το stress test θα είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε αν αυτά λειτουργούν σωστά. Ε, σήμερα δε, ε, δεν έχω ψευδεστήσεις για το τι υπάρχει. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά ε, το δισταγμό με τον οποίο προχωρά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και αν δεν έχουμε μία συντονισμένη διαδικασία δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε ίσως όχι την επόμενη κρίση αλλά τα δυνητικά προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να σας καθυστερήσω, λέει ο κύριος Μπούλμαν και γι' αυτό μιλάω αγγλικά. Αλλά θα υπάρχουν επικερδείς συζητήσεις. Το ερώτημα ήταν τι μαθήματα αποκομίζουμε από την κρίση κατά τρόπον ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο για τη συμπεριφορά των βασικών ε, εμπλεκομένων διότι λέμε να ακούσουμε τα, τις αγορές, να ακούσουμε τα κράτη-μέρη, να είμαστε φιλόδοξοι αλλά εγώ ρωτώ εσείς τι μπορείτε να συμβάλλετε κατά τρόπον ώστε να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση με παρακολούθηση των πράξεων των βασικών εμπλεκομένων. Με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι η ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν συνεργαστεί σε πολλά θέματα με καλή έκβαση. Αυτό που θεωρώ βασικό είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και τη συνεργασία και να την ενισχύσουμε κατά τρόπον ώστε οι φιλοδοξίες και οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιτευχθούν. Απαντώ στην ερώτησή σας, γιατί αν όχι ε, δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Είμαι βέβαιος και προσβλέπω στο να το ξανασυζητήσουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία και ελπίζω ότι θα, το, θα τα ξαναπούμε από αυτού. Η μέθοδος έχει σημασία, αλλά η ουσία είναι διαφορετική και γι' αυτό διαφέρουμε. Κυρία Φόρντ, γενικά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα θέμα σχετικά με τη Βασιλεία 3. Τώρα σας βλέπω. Ναι, είπα όντως ε, αυτό το σχόλιο αλλά είπα ότι η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για την πλήρη και συνεκτική εφαρμογή της Βασιλείας 3. Εάν οι δύο ε, δικαιοδοσίες αποτύχουν ο υπόλοιπος κόσμος δεν πρόκειται να εφαρμόσει αυτή την ρύθμιση. Δεύτερον, είπα κάτι στους τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες συνεχίζουν να παραπονούνται γιατί θέλουν να υπάρχει ισοτιμία όσον αφορά τις ενέργειες. Εσείς λέτε ότι οι Ευρωπαίοι τραπεζίτες εξαιρούνται από τη Βασιλεία 3 και το ίδιο λένε άλλοι τραπεζίτες και προσπαθούν να αποδυναμώσουν την Βασιλεία 3 μέσα στο δικό τους εθνικό χώρο. Άρα όλοι αυτοί φέρουν ευθύνε. Αυτό ήθελα να πω. Σχετικά με την ευελιξία για να είμαστε πιο αυστηρή από τις προϋποθέσεις της Βασιλείας 3 πιστεύαμε πάντοτε ότι η Βασιλεία 3 θα ήταν η ελάχιστη προϋπόθεση για το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα. Βλέπουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλοι συνεργαζόμαστε. Άρα χρειάζεται αμοιβαία εξήγηση και διαφάνεια ε, μεταξύ μας. Τώρα ο Ζων Πολ. Θα είσαι ο πρώτος. Του επόμενου γύρου. Ορίστε Ζων Πολ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Διοικητά. Θα είστε λοιπόν πρόεδρος του FSB. Η κρίση των χρεών που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα στοιχείο του συστημικού κινδύνου. Τι θεωρείτε λοιπόν ότι με βάση τις παρατηρήσεις σας είναι άλλοι πιθανοί λόγοι συστημικών κινδύνων που πρέπει να προσέξετε. Α, σύντομα το ερώτημα, αλλά θα υπάρξουν σίγουρα και άλλα. Κύριε ε, Δικητά, κύριε υποψήφιε, εγώ έχω μία ερώτηση που αφορά στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου και μία σχέση με την με το Επιστημονικό του Συμβούλιο. Αποφασίσαμε να συσταθεί αυτό το Επιστημονικό Συμβούλιο, το άρθρο 12.3 του κανονισμού για την, Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου ε, προβλέπει ότι το Συμβούλιο αυτό μετά από εντολή του διοικητή ή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δραστηριοποιείται. Αυτό σας αφορά δηλαδή. Και τι θέλω να ρωτήσω. Αυτό το επιστημονικό συμβούλιο θα του αναθέσετε μία, θα μία ευρεία εντολή έτσι ώστε μόνο του να μπορεί να λειτουργεί, ε, να λειτουργεί αυτεπάγγελτα χωρίς να περιμένει εντολές από εσά να αναλαμβάνει μόνο του ε, πρωτοβουλίες. Επίσης θα μεριμνήσετε έτσι ώστε αυτό το Συμβούλιο να δημοσιοποιεί τα πορίσματά του στο βαθμό βέβαια που κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο. Ο κύριος Κλούτ, Γιώργεν Κλούτ. Οι, δική μου, οι δικές μου ερωτήσεις καλύφθηκαν και επειδή δεν υπάρχει χρόνος παρετούμε. Δεν θέλω να κάνω άλλη ερώτηση. Κύριε Ντράγκη, σας προσφέρω το χρόνο μου για να απαντήσετε. Πολύ ωραία. Και η τελευταία ερώτηση ε, από την Κλόντια Μακάμπλη. Eh, σας ευχαριστώ ε, κύριε Ντράγκη που ήρθατε εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ. Ε, μία ερώτηση αφορά ε, στους οίκους αξιολόγησης. Αυτοί είναι οργανισμοί που έχουν τεράστια εξουσία, ανεξέλεγκτη εξουσία στις διεθνείς αγορές και θέλω να ακούσω τη δική σας τη γνώμη γιατί τρεις αμερικανικοί οίκοι αξιολόγηση ελέγχουν το σύνολο της αγοράς και κάνουν τεράστια λάθη. Αναφέρεται προηγουμένω στην περίπτωση της Lehman Brothers αλλά για αυτή την περίπτωση δεν υπέστησαν τις συνέπειες που έπρεπε προκαλούν ζημιές, ε, έλλειψη ισορροπίας σε χώρες με λάθος εκτιμήσεις τους. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ψήφισε ένα ψήφισμα που ζητάει μεγαλύτερες ε, ευθύνες, λογοδοσία σε αυτό τον τομέα. Η δική σας άποψη ποια είναι και τι είδους πρωτοβουλίες έχετε να προτείνετε έτσι ώστε να υπάρχει πράγματι διαφάνεια και ανάληψη ευθυνών. Και μια άλλη ερώτηση. Μιλήσαμε πολύ σήμερα για χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία υπήρχαν κάποιες ενδείξεις δυσκολίες κατά παρελθόν. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις ε, ε, ως πρόεδρος ε, της ΕΚΤΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου θα δράσετε στο μέλλον, θα θελήσετε να λάβετε κάποια πρωτοβουλία για να προλάβετε κάποιες καταστάσεις. Right. So that's the final round of questions. Μάλιστα. Τελευταίος γύρος τελείωσε, ορίστε. Ευχαριστώ. Κύριε Κοζές Για να σας απαντήσω. Θα έπρεπε να αναφέρω ποιοι είναι οι συστημικοί παράγοντες σε αυτή τη συγκυρία και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Είναι ερώτημα που, που αφορά τελικά τι εκκρεμεί ακόμα στη μεταρρύθμιση του συστήματός μας, του δημοσιονομικού μας συστήματος. Το πρώτο θέμα που πρέπει να δούμε αφορά αυτά που είπα πριν, δηλαδή απαντώντας στην κυρία Φόρο, ότι δηλαδή πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Βασιλεία 3 θα εφαρμοστεί πλήρως και μάλιστα με συνεπή τρόπο παγκοσμίω. Υψηλότερα κεφάλαια και καλύτερης ποιότητας. Οι κανόνες για τη ρευστότητα δεν έχουν ακόμη πλήρως εξεταστεί, αλλά θα χρειαστεί να εφαρμοστούν όταν θα έχει τελειώσει η λεγόμενη αξιολόγηση, μελέτη αξιολόγησης. Η... Ύστερα πρέπει να δούμε τι ευθύνεται περισσότερο από τι άλλο για τους ηθικούς για να το πω έτσι κινδύνους. Τρεις ιδέες εδώ κυριαρχούν. Πρώτον περισσότερα κεφάλαια. Ακόμη περισσότερα από ό,τι για τις υπόλοιπες τράπεζες σε εκείνες που εμπεριέχουν κινδύνους. Και δεύτερον το κυριότερο και το πιο δύσκολο ένα σύστημα που να μπορεί να διαχειρίζεται μεγάλες αποτυχίες χωρίς να χρειάζεται να τις πληρώνει ο, καταναλω... φορολογούμενος και χωρίς να διαταράσσονται οι αγορές. Η Κομισιόν προετοιμάζει μια σχετική πρόταση που την αναμένω και εγώ. Σε τρεις φάσεις την προετοιμάζει. Πρέπει να περιορίσουμε την εθνική ευχέρεια σε αυτό, για αυτό το πρόβλημα γιατί μερικά προβλήματα μόνο σε ενωσιακό πλαίσιο μπορούν να λυθούν. Πώς θα διαχειριστούμε λοιπόν μία αποτυχία, ποιοι πιστωτές θα προστατευθούν, ποιοι θα ωφεληθούν από κάποια πτώχευση ή αποτυχία. Και τρίτη μέθοδος, πώς θα μπορούσαν οι επιτηρητές, οι επόπτες να είναι πιο ανεξάρτητοι πιο ισχυρή έναντι των μεγάλων τραπεζών. Μερικές φορές μάλιστα ε, και των κυβερνήσεων, γιατί μερικές φορές οι επόπτες εξαρτώνται από κυβερνήσεις. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία και των εποπτών και των τραπεζών, κεντρικών τουλάχιστον, γιατί μπορεί εδώ να υπάρξουν κοινά συμφέροντα με τις ιδιωτικές τράπεζες. Πρέπει να μειωθεί ο ηθικός κίνδυνος που εμπεριέχει η λειτουργία αυτών των μεγάλων οργανώσεων. Άλλη ιδέα είναι η λεγόμενη σκιώδης τραπεζική δραστηριότητα, shadow banking, γιατί πρέπει με βαθύτερο, ισχυρότερο τρόπο να διευθετήσουμε, να διαχειριστούμε τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Αλλά υπάρχουν δραστηριότητες που γίνονται λίγο πολύ κρυφά στη σκιά το πρώτο που θα έπρεπε να δούμε είναι να δούμε τι εύρος έχει αυτή η μη παράνομη δραστηριότητα. Και η απάντηση είναι θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε σε οτιδήποτε σε αυτές τις δραστηριότητες εμπεριέχει δανειοδότηση, δανεισμό. Αν κάποιος δηλαδή δρά ως τράπεζα, ακόμη και αν δεν λέγεται τράπεζα, θα πρέπει να του εφαρμόζονται οι ίδιοι κανονισμοί όπως στις τράπεζες. Οι ίδιοι κίνδυνοι, ε, τότε και η ίδια νομοθεσία, οι ίδιοι κανόνες. Έτσι θα λύσουμε το θέμα της των σκιωδών τραπεζών. Ε, rightly, many people said that... Τέλος, το θέμα των OTC derivatives που είναι κύριος τρόπος διεύρυνσης των κινδύνων. Θυμηθείτε τι έγινε με τους Lehman Brothers. Δεν ξέραμε ούτε καν το εύρος των δραστηριοτήτων τους εκεί. Ακούγονταν αριθμοί που κάθε μέρα άλλαζαν και δεν ξέραμε τι ακριβώς έκαναν. Πρέπει λοιπόν πρώτα πρώτα να γνωρίζουμε περισσότερα να υπάρξει ένας συγκεντρωτισμός των παραγόγων, να λέμε ότι τα παράγωγα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε κεντρικά από κεντρικούς οργανισμούς για να γνωρίζουμε ποιος είναι από πίσω, πόσο κεφάλαιο διαθέτει και πώς το διαχειρίζονται. Αυτές τις πληροφορίες δεν τις είχαμε το 8 και το 9. Ποιες εγγυήσεις έχει. Λοιπόν, τα παράγωγα αυτά θα τα χειριζόμαστε αυτά που δεν μπορούν να τύχουν τέτοια συγκέντρωση δηλαδή και γι' αυτά πρέπει να γίνει κάτι. Θα χρειάζεται τουλάχιστον να καταθέτουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούμε σε ειδικά ιδρύματα που θα λέγονται trade repositories και θα υπάρχει πρόσβαση των δημοσίων αρχών σε αυτές τις πληροφορίες. Αυτή είναι η κύριοι τομείς όπου πρέπει να προσπαθήσουμε τους επόμενους μήνες να διευθετήσουμε τα πράγματα. Και θα γίνουν προτάσεις τον Νοέμβριο στο Παρίσι στη συγκέντρωση του G20. Αλλά και τα επόμενα χρόνια πρέπει να γίνει κάτι. Ο δρόμος είναι καθαρός λοιπόν. Ξέρουμε που θέλουμε να πάμε και με τη στήριξη που είχαμε μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε επενδεδημένα συμφέροντα αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ ενεργά, πολύ δραστήρια. Μέχρι τώρα δεν είχαμε πλήρη αποτυχία μπορώ να πω σε αυτό. για το ανεξάρτητο συμβουλευτικό σώμα ή ακαδημαϊκό σώμα που αναφέρατε. Γι' αυτό το θέμα λέω συχνά ότι η αξία της ύπαρξης ενός τέτοιου επιστημονικού συμβουλίου είναι, έγκυται ακριβώς στην ανεξαρτησία του. Απαντώ λοιπόν ότι θα πρέπει τις συμβουλές του να τις δίνει ανεξαρτήτως, με ανεξάρτητο τρόπο. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά όλα όσα είπατε για το ανεξάρτητο συμβουλευτικό συμβούλιο που πρέπει να δρά και ανεξάρτητα είπατε. Θα μιλήσω αγγλικά, ίσως ε, αυτό είναι πιο σαφές. Και τελικά στην Ευρώπη θα μιλάμε όλοι αγγλικά. Η ερώτηση είναι εξής με βάση το άρθρο 12.3. Αναφέρεται στο άρθρο αυτό του κανονισμού με απόλυτη σαφήνεια ότι το Συμβούλιο αυτό δραστηριοποιείται μετά από αίτημα του Πρόεδρου. Άρα δηλαδή εσείς ως ε, επίδοξος Πρόεδρος μπορείτε να μας πείτε τώρα τι θα κάνετε. Θα δώσετε εντολή στο Συμβούλιο να επεξεργάζεται μόνο του τα δικά του θέματα. Θα δίνει συμβουλές στην ESRB και εν πάση περιπτώσει θα τους επιτρέπετε ε, να δημοσιεύουν τα πορίσματά τους, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο. Κοιτάξτε, ε, μικροδιαχείριση δεν είναι το δικό μου το στυλ. Εγώ είμαι ακαδημαϊκός, ε, προέρχομαι από τον ακαδημαϊκό χώρο και ξέρω πόσο χρήσιμη είναι η ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Όπως σας είπα, ε, το Συμβούλιο αυτό θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητο, αλλιώς δεν το χρειαζόμαστε. Όσον αφορά τώρα τις δημοσιεύσεις, αυτή είναι μια συλλογική απόφαση. Θα πρέπει να αποφασίσουμε περισσότερο γι' αυτό. Δεν το αποκλείω, αλλά θα πρέπει βέβαια να ακούσω και την άποψη των υπολείπων μελών ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της ESRB, τι έχουν να πούν αυτοί επ' αυτού. Κύριος μοργκάντη. Απευθύνομαι στον κύριο μοργκάντη. Τώρα, όσον αφορά τους ε, οίκους αξιολόγησης, η εμπειρία μας μέχρι τώρα είναι ότι πράγματι οι και αυτοί ε, επικρίθηκαν δρυμύτατα κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση και λήφθησαν αρκετά μέτρα στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη για να αντιμετωπιστούν οι πλέον κατάφορες ε, παραβιάσεις συμφερόντων, συγκρού συμφερόντων που εντοπίστηκαν σε οικου αξιολόγηση. Τώρα λοιπόν έχει διασφαλιστεί πλέον μεγαλύτερη διαφάνεια, ε, πλήρη διαχωρισμό ανάμεσα στο rating και στην παροχή συμβουλών, στην αξιολόγηση και την παροχή συμβουλών, δύο ξεχωριστά πράγματα. Έχουμε ένα πρόγραμμα του πώς θα μπορέσουμε ίσως ε, να ξεφορτωθούμε κατά λέξη αυτούς τους οίκους αξιολόγησης. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση επ' αυτού. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Πρώτον τους ρυθμιστές, κατόπιν τους επενδυτές και τρίτον issuers, όσοι κάνουν τις εκδόσεις. Όσον όπως ξέρετε, όσον αφορά τους ρυθμιστές, ε, ε, πολλοί δεν ε, συμπεριλαμβάνουν τις αξιολογήσεις του στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Βασιλεία 3 ε, χρησιμοποιεί την αξιολόγηση CRE για την αξιολόγηση κινδύνων που απειλούν τις τράπεζες. Αυτό όμως δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να μετράτε ο κίνδυνος. Το ίδιο ισχύει και για τις εγγύησεις που εκδίδει η ΕΚΤ. Τους λέμε, εντάξει, να δούμε λίγο τις αξιολογήσεις των οίκων αυτών αλλά πρέπει και μόνοι μας να αξιολογήσουμε τους ε, κινδύνους ε, των ε, διαφόρων τραπεζών. Θέλω να πω λοιπόν το εξή, ότι ο τελικός στόχος είναι να αποφασίσει κανείς μόνος του το τι συνιστά κίνδυνο και τι όχι. Και κατά πόσον ομόλογα ενέχουν κινδύνου ή όχι. Πάνω δεν υπάρχει απόλυτη αντικειμενικότητα. Αυτό το βιώσαμε και με τους επενδυτές. Μάλιστα, ε, προς έκπληξή μας ε, διαπιστώσαμε, οι θεσμικοί επενδυτές είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τη γνώμη των οίκων αξιολόγησης. Γιατί πολλές φορές μόνοι τους, ε, στους θεσμούς τους μέσα, δεν έχουν επιτροπές για να αξιολογήσουν τους κινδύνους. Εύκολη λύση λοιπόν να καταφεύγουν στην άποψη των οίκων αξιολόγησης, έστω και αν αυτή είναι ατελής. Στόχος μας λοιπόν ως ρυθμιστές είναι να χρησιμοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δική μας την αξιολόγηση κινδύνων. Δεν είναι εύκολο αυτό να εφαρμοστεί, αλλά ξέρουμε ε, πού πρέπει να κατευθυνθούμε. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο κύκλος των ε, ερωταπαντήσεων και δεν είναι απαραίτητο να κάνετε μια καταληκτική ε, ομιλία, ένα σχόλιο, αλλά αν κρίνετε ότι κάτι δεν ελέγχθησε αυτές τις μισή ώρες, τώρα έχει την ευκαιρία να το πείτε. Θα είμαι πολύ σύντομος, διότι είναι η πρώτη μου εμπειρία να είμαι δημοκρατικά υπόλογος. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και για μένα ήταν ε, πολύ διδακτική και γι' αυτό και εδώ και πολύ καιρό ήθελα να έρθω. Σας είμαι ευγνώμων για όλες τις ερωτήσεις τις οποίες μου απευθύνεται και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ελπίζουμε αν όλα πάνε καλά θα έρχεστε εδώ έξι φορές το χρόνο. Θα γνωριστούμε λοιπόν πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα, η διαδικασία είναι η εξής τώρα ότι πρέπει να φύγουν όλοι εκτός των Ευρωβουλευτών και των βοηθών βεβαίως Δηλαδή θα κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα για να μπορέσουν οι πολιτικές ομάδες να συζητήσουν μεταξύ τους προτού συνεχίσουμε με μια ανοιχτή συζήτηση.